afternoon, ladies uh, Καλησπέρα σας ε, κυρίες και κύριοι παρακαλώ καθίστε για να ξεκινήσουμε αντικαθιστώ σήμερα τον κύριο Λάγκε, τον πρόεδρό μα, ο οποίος ε, δυστυχώς κολλείεται έχετε την ημερήσια διάταξη. Υπάρχει κάποια αντίρρηση ή εγκρίνεται. Δεν βλέπω κάποια αντίρρηση. Οπότε εγκρίνεται. Ωραία. Λοιπόν, έρχομαι στις δύο ανακοινώσεις ε, του Πρόεδρου. Όπως ξέρετε, η συνεδρίαση μας ως συνήθως μεταδίδεται. και θα ήθελα να σας παρακαλέσω λόγω της ερμηνείας να μην μιλάτε πάρα πολύ γρήγορα. Σημείο 3. Αποφάσεις των συντονιστών. Συνεδρίασαν οι συντονιστές στις 18 Ιουλίου και βεβαίω ε, οι αποφάσεις του αφορούν τη σημερινή ημερήσια διάταξη. Θα ήθελα να αναφέρω κάποιες από τις αποφάσει, δηλαδή την απο... η γνωμοδότηση για τον προπολογισμό του 2020 θα είναι υπομορφή επιστολής ε, και δόθηκε στον πρόεδρο τη Επιτροπή, τον κύριο Μπέρντ Λάγκε. Ε, κατά τα λοιπά, ε, άλλες αποφάσεις θα περιληφθούν στα πρακτικά της ε, σημερινής συνεδρίασης για, μια... για να εγκριθούν σε μια συνεδρίαση του Σεπτεμβρίου. Αυτά όσον αφορά τα πιο τυπικά και τώρα περνάμε στην παρουσίαση της Επιτρόπου Μάλμστρομ την οποία θα ήθελα να ευχαριστήσω για την ευελιξία της, γιατί ξέρετε ότι λόγω τεχνικών λόγων ακυρώθηκε η πτήση της σήμερα το πρωί. Πρέπει να πάρει άλλη πτήση. Ευχαριστώ και εσάς για την ευελιξία σας, γιατί τελευταία στιγμή ειδοποιηθήκατε ότι άλλαξε το χρονοδιάγραμμα. και αλλάξατε το πρόγραμμά σας ε, για να έρθετε εδώ. Έχουμε αρκετά μεγάλη προσέλευση. Σας ευχαριστώ λοιπόν για την ευελιξία που επιδείξατε. Σας ευχαριστώ κυρία Επίτροπε. Η ανταλλαγή απόψεων για τις τελευταίες εξελίξεις ε, είναι κάτι το οποίο αναμένουμε. Εν τω μεταξύ, είχαμε δύο σημαντικές εξελίξεις. Η μία ήταν ότι μετά από 20 χρόνια διαπραγματεύσεων επετεύχθη μια συμφωνία επί της ε, αρχής ε, με τις χώρες της ε, Μερικοσούρ, Αργεντινή, Βραζιλία, Παραγουάι, Ρουάι και αυτό σημαίνει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα είναι πλέον εμπορικός εταίρος των χωρών αυτών και θα μιλάμε για τη μεγαλύτερη εμπορική συμφωνία που έχει συνάψει ποτέ η Ένωση. Μέχρι τώρα μεγαλύτερη τέτοια συμφωνία ήταν αυτή με την Ιαπωνία, τώρα θα αντικατασταθεί από αυτήν με το Μερκοσούρ. Βεβαίως είχαμε αρκετές ε, εντάσεις ε, και θα, μα θα μας εξηγήσει η κυρία Επίτροπος δύο μέρες αργότερα στις 13 Ιουλίου υπογράψαμε μια εμπορική συμφωνία και συμφωνία επενδύσεων με το Βιετνάμ θα θυμάστε ότι έχουμε ξανά υπογράψει στο παρελθόν αλλά λόγω της απόφασης του ΔΕΚ έπρεπε να την επαναδιαπραγματευτούμε και να σπάσουν σε δύο κομμάτια αυτές οι συμφωνίες, ένα κομμάτι εμπορική και ένα κομμάτι επενδυτική. Υπογράφηκαν και τα δύο και τέλος. Προετοιμαζόμαστε για την διαδικασία σύμφωνης ε, γνώμης επί των συμφωνίων αυτών και υπάρχουν και άλλα ζητήματα που θα μας απασχολήσουν. δεδομένου των τελευταίων εξελίξεων στις σχέσεις με τις ΗΠΑ. Κάνατε κάποιες παρατηρήσεις για τις διαπραγματεύσεις με Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία, οπότε είμαστε στην διάθεσή σας για να ακούσουμε. Και μετά να κάνουμε τις παρατηρήσεις μας. Έχετε τον λόγο κυρία Επίτροπε. Ευχαριστώ Πρόεδρε, καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Σας ευχαριστώ για την ευελιξία σας. Είχα φρικτό πρωινό καθυστερημένες ακυρωθήσεις πτήσεις. Σας ευχαριστώ που ήσασταν ευέλικτοι. έβλεπα στη συνάντηση μαζί σας. Συγχαρητήρια στους νεκρογέντες και νεκλογήσεις. Παραδοσιακά έχουμε καλή συνεργασία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αυτή η Επιτροπή και παρά το σύντομο εναπομένο χρονικό διάστημα ελπίζω να συνεχιστεί. Τα εμπορικά θέματα και άλλωστε γι' αυτό επιλέξατε να είστε αυτή την Επιτροπή, είναι πολύ επίκαιρα αυτές τις μέρες. Έχουμε διαφορετικές σε διαφορετικές τάσεις εμπορικούς πολέμους, μονόπλευρες δράσεις που στέφονται κάτω κανόν του ΠΟΕ, απειλές κατά του ΠΟΕ και πολλές συγκρούσεις. Συζητήσεις με τη ΣΥΠΑ, με την Κίνα, έχουμε ένα κράμα πολιτικής ασφαλείας με δασμούς, κάτι που δεν είδαμε ποτέ πριν. Άρα πολλά προσυζήτηση στον εμπορικό τομέα Ευρωπαϊκή Ένωση με την ισχυρή υποστήριξη αυτής της Επιτροπής προσπάθησε στην προηγούμενη θητεία να τοποθετηθεί εντός όλων αυτών ούτως ώστε η εμπορική πολιτική να είναι ανοιχτή, να καλύπτει όλους, να είναι διαφανής, να βασίζεται επί αξιών και να εστιάζουμε περισσότερο στην υλοποίηση, επιβολή και παρακολούθηση. Συνεργαζόμαστε με φίλους μας, έχουμε σε επαφή μαζί τους πολυμερώς για να εξυγχρονίζουμε, να μεταρρυθμίζουμε τον ΠΟΕ και συνεργαζόμαστε με τον κύκλο φίλων, διμερός ή περιφερειακός, ούτως ώστε να δημιουργήσουμε ένα δίκτυο. Δίκτυο χωρών που έχουν τις ίδιες με μας, πιστεύουν στο προοδευτικό εμπόριο που βασίζεται σε αξίες, αλλά που εδράζεται επί του πολυμερού συστήματος διότι πιστεύουμε ότι πρέπει να εμπορευόμεθα ένας με τον άλλον, είναι αμοιβαία εποφελές αν είναι βιώσιμο το εμπόριο, αν λειτουργεί σωστά και αν εδράζεται επί πολυμερών αρχών. Γι' αυτό συνάψαμε συμφωνία τώρα με τον Καναδά, την Ιαπωνία, με τη Σιγκαπούρη, με το Μεξικό. Στην τελευταία φάση λεπτομέρειε ρυθμίζουμε για τι κρατικέ προμήθειε με τη Χιλή, τη Νέα Ζηλανδία, την Αυστραλία και την Ινδονησία και όπως είπε και ο Πρόεδρος, πρόσφατα υπογράψαμε με το Βιετνάμ. Από εσά εξαρτάται τώρα να προωθήσετε το θέμα και μετά από 20 χρόνια τελειώσαμε διαπραγματεύσεις με τέσσερις χώρες του Μέρκοσουρ. Αν επιτρέπετε, Πρόεδρε, θα ήθελα να αναφερθώ στις δύο συμφωνίες, Βιετνάμ και Μερκοσούρ. Αναφέρα και τον είπα και την κατάσταση στον ΠΟΕ. Μπορώ να απαντήσω σε σχετικές ερωτήσεις ό,τι αφορά το εμπόριο αλλά να αφήσω και κάποιο χρονικό διάστημα για ερωτήσεις. Μερκοσούρ λοιπόν, 28 Ιουνίου, η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Μερκοσούρ κατέληξαν σε μια πολιτική συμφωνία που είναι ισορροπημένη, φιλόδοξη, πλήρης συμφωνία εμπορική, που αποτελεί και ένα τμήμα συμφωνίας σύνδεση και εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο συνεργασία. Είναι ύψη τη γεωπολιτική σημασία, όπω καταλαβαίνετε, με φίλου και συμμάχους στη Λατινική Αμερική που έχουμε μακρά ιστορία επαφής μαζί τους και πολιτισμικής συμμαχίας και στέλνουμε ένα ισχυρό μήνυμα για διεθνές εμπόριο που βασίζεται σε κανόνες και σχέσεις που είναι προβλέψιμες και συμφωνίες που είναι προβλέψιμες διεθνείς. Είναι από πλευρά εμπορικών πολιτικών καλή συμφωνία, θα δώσει στι ευρωπαϊκέ επιχειρήσει σημαντικό προβάδισμα σε μια μεγάλη αγορά με μεγάλη δυνατότητα για ανάπτυξη. Για τα εγαθά το Mercosur έρει τα τέλη για 91% των προϊόντων που εισάγονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είμαστε η πρώτη οικονομική δύναμη που συνάπτει εμπορική συμφωνία με τη Mercosur. Έχουμε το όφελο εκείνο που πρώτο κινείται σε αυτήν την αγορά. Πάνω από 260 εκατομμύρια καταναλωτέ βρίσκονται εκεί. Και από πλευρά δασμών θα έχουμε οικονομίε ευρωπαϊκή επιχειρήσει 4 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο, 8 φορέ όσο με τον Καναδά και, όσο και 4 φορέ όσο η Ιαπωνία και ανοίγει πρόσβαση για παροχή υπηρεσία, κρατικών προμηθειών, θαλασσίων μεταφορών και υπηρεσιών σε μια περιοχή που θα επενδύσει πάρα πολλά σε σύγχρονε υποδομέ. Κάποιοι θα το αφισβητήσετε, αλλά λέω ότι είναι μια καλή συμφωνία για του γεωργού μα. Έχουμε προϊόντα υψηλή προθυμισταξία όπω είναι το τυρί, το κρασί, το ελαιόλαδο, τα λαχανικά, όπως και κονσερβασμένα προϊόντα, όπως είναι γλυκά, όπως είναι ε, σοκολάτα κλπ. Να βάλουμε υπόψη διάφορε ευαισθησίε όπου εκείνα τα προϊόντα όπω είναι το βόλιο κρέα, η ζάχαρη και τα πουλερικά μέσω προσεκτική σταθμισμένη ε, ποσόστοσης και δασμών θα περιορίζονται σε όγκο και επί σειρά ετών σταδιακά θα αυξάνεται. Λοιπόν, είναι μόνο ένα μικρό ποσοστό, το 1% ε, τα πουλερικά, το χείριο κρέας στις αγωγέ και το βόλιο. Έχουμε μηχανισμό διαφύλαξης και εμείς και οι τέσσερι χώρε Μερικοσούρ μπορούμε προσωρινά να επιβάλλουμε προσωρινά μέτρα για να ρυθμίσουμε εισαγωγέ σε περίπτωση απροσδόκητων σημαντικών αυξήσεων στι εισαγωγέ που μπορούν να δημιουργήσουν, να απειλήσουν, να δημιουργήσουν σοβαρή ζημιά στι εσωτερικέ αγορέ. Η συμφωνία προστατεύει πάνω από 350 ενδείξεις προέλευση για ΡΗ, είναι ο πνευματόδη της Ευρώπης και την ίδια προστασία θα χαίρουν όπως και εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυτά τα προϊόντα και είναι μεγάλη νίκη για τη γεωργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτό. Επίσης είναι μια συμφωνία που προωθεί τις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει φιλόδοξο κεφάλαιο που αναφέρεται στη βιώσιμη ανάπτυξη, δεσμεύονται και τα δύο μέρη να σέβονται τις διεθνείς κανόνες και τις συμφωνίες για το περιβάλλον, καλύπτεται η βιώσιμη διαχείριση και η συντήρηση των δασών, το σεβασμό των εργασιακών δικαιωμάτων και ε, επίση η ε, υπευθυνότητα των επιχειρήσεων προωθείται. Θα πρέπει τα μέρη, τα συμβαλόμενα, να εφαρμόζουν αποτελεσματικά διάφορε υποχρεώσει που λαμβάνονται στι συμβάσει του Διεθνού Γραφείου ε, Εργασία και έχουμε κεφάλαια βιώσιμη ανάπτυξη και συμφωνούν τα συμβαλόμενα μέρη να εφαρμόζουν αποτελεσματικά διεθνεί συμβάσει για το περιβάλλον και να καταπολεμήσουν το παράνομο εμπόριο, κυρίω τα αγρια ζώα. Ενθαρρύνεται επίση η εμπορία προϊόντων που αποκτούνται από βιώσιμα διαχειριζόμενα δάση και χρειάζεται οι ηθαγενείς πρώτα να συμφωνήσουν και οι τοπικές κοινότητες που ε, κατοικούν στα δάση. Στη συμφωνία και οι δύο εταίροι, εμείς και οι χώρες Μερκοσούρ δεσμευόμεθα αποτελεσματικά να εφαρμόζουμε τη Συμφωνία των Παρισίων για την αλλαγή του κλίματος. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε δεσμευτεί να καταπολεμήσουμε την αλλαγή του κλίματος και να συνεργαστούμε προς μια μετάβαση προς μια οικονομία που θα είναι χαμηλή σε άνθρακα. Αυτό είναι σημαντικό, διότι έτσι οι υποχρεώσει μα που έχουν αναλυφθεί ε, στην Συμφωνία των Παρισίων ότι Υπάρχουν δυνάμει στον κόσμο που θα ήθελαν να ακολουθήσουν διαφορετική πορεία, να αποσυρθούν από τη Συμφωνία των Παρισίων, αλλά εδώ στηρίζουμε, δένουμε τους τέσσερις εταίρου μα το Μερκοσούρ με τη Συμφωνία των Παρισίων, με ε, νομικά δεσμευτικέ υποχρεώσει και έχουμε και μηχανισμό διευθέτησης ε, διαφορών διατηρούμε το δικαίωμα να ρυθμίζουμε τις δημόσιες ε, προμήθειες και τα πρότυπά μας στον φυτογειονομικό τομέα. Όλα αυτά διαφυλάσσονται πλήρως. Υπάρχει αναφορά στην αρχή της πρόληψης και τίποτα σε αυτή τη συμφωνία δεν αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο εμείς υιοθετούμε και εφαρμόζουμε ε, τους κανόνες περί της υγιεινής των τροφίμων. Είτε αυτά παράγονται τοπικά είτε εισάγονται τα τρόφιμα. Επίσης θέλουμε να προωθήσουμε τις αξίες για την επαφή με τους εμπλεκόμενους φορείς, κοινωνικό διάλογο, συνεργασία με την κοινωνία των πολιτών που πρέπει να συμμετέχει ενεργά στην εφαρμογή των κανόνων και να συζητούμε με του εταίρους μα για θέματα περιβαλλοντικά και σχετικέ ανησυχίες. Όπως θα είδατε, η πλήρη συμφωνία πέρα από κάποια τμήματα του IPR, του κεφαλαίου IPR, όπου εκεί προσπαθούμε να χτενίσουμε το κείμενο για λεπτομέρειε, δημοσιεύτηκε 12 Ιουλίου από όταν ολοκληρώθηκε οι διαπραγματεύσει με το Mercosur, τα κείμενα δημοσιεύθηκαν ταχύτερα από οποιαδήποτε άλλη συμφωνία. Εν τω μεταξύ, στην προηγούμενη θητεία είχαμε τακτικές επαφές με αυτή την επιτροπή, την επιτροπή σας και με την ομάδα την αρμόδια. Και η κυρία Γκαλίνη, επικεφαλή επικεφαλής διαπραγματεύτρια, ήταν εδώ για να απαντήσει στα μέλη του Κοινοβουλίου. Τώρα ε, αναθεωρούμε νομικά το κείμενο, ε, το χτενίζουμε νομικά και μετά θα μεταφραστεί σε όλες τις γλώσσες το κείμενο αυτό και μετά εξαρτάται από το Συμβούλιο και μετά θα έρθει στα χέρια σας. Αλλά υπάρχουν ακόμα κάποια χρονικά περιθώρια, όχι φτάσουμε εκεί, έχετε χρόνο να εξετάσετε, να συζητήσετε το θέμα και οι συνεργάτες μου και εγώ στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή με τα χαράς να συζητήσουμε πάνω σε αυτά τα θέματα. Τώρα, όσον αφορά το Βιετνάμ, όπω είπε και ο Προέδρο, στις 30 Ιουνίου υπεγράφει η Συμφωνία Ελευθέρου Εμπορίου και η συμφωνία για την προστασία των επενδύσεων στο ΑΝΟ. Οι δύο συμφωνίε είναι σημαντικό βήμα για την ενίσχυση των διμερών μα σχέσεων μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωση και Βιετνάμ, βασιζόμενοι σε ε, ήδη δεσμού στενού που είχαμε στον τομέα του εμπορίου και των επενδύσεων. Τώρα θέλαμε ανθρώπινα δικαιώματα, εργασιακά δικαιώματα να προστατεύονται και το περιβάλλον και έτσι θα δώσουμε και άλλα στοιχεία του πόσο αφοσιωμένοι είμαστε εμεί ε, στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Ασία επιβεβαιώνει η δέσμευσή μας να ανοίξουμε το εμπόριο να είναι δίκαιο εμπόριο. Έχουμε πολλέ φιλοδοξίε όσον αφορά την πρόσφυση στην αγορά για αγαθά υπηρεσίε και προμήθειε, για κανόνε και ε, γεωγραφικέ ενδείξει, διευκόλυνση των τελωνιακών διαδικασιών και τεχνικού φραγμού, τεχνικού στο εμπόριο. Πρέπει να έρθουν. Το πεδίο εφαρμογή. Το πλαίσιο απελευθερώνει περίπου 99% τη εμπορία αγαθά. Αυτό είναι κάτι άνευ προηγουμένου σε μια αναπτυσσόμενη χώρα Οπότε στέλνουμε σημαντικότατο μήνυμα και είναι ένα σημείο αναφορά αυτό για μελλοντικέ συμφωνίε με άλλου εταίρους ε, στην ε, περιοχή. Συμπεριλαμβάνονται δεσμεύσει για την προστασία των δικαιωμάτων εργαζομένων, το σεβασμό των βασικών προτύπων εργασία του ILO και κύρωση των σχετικών συμβάσεων. Και ξέρω ότι αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για την Επιτροπή σα. Το Βιετνάμ πριν από δύο εβδομάδε περίπου κύρωσε μία από τι τρει εκκρεμούσε συμβάσει του ILO και έχει επιβεβαιώσει χρονοδιάγραμμα σε μια επιστολή που διαβίβασα στην Επιτροπή για τις δύο αναπομένουσες συμβάσεις και θα υιοθετήσει αναθεωρημένο κώδικα εργασιακό ε, το φθινόπωρο, αργά στο φθινόπωρο και αυτό δεν θα είχε συμβεί χωρίς αυτή τη συμφωνία για το ελεύθερο εμπόριο. Η συμφωνία επίσης συμπεριλαμβάνει δεσμευτικές υποχρεώσεις για το περιβάλλον, προστασία του περιβάλλοντος, συμφωνία των Παρισίων, το ε, πρωτόκολλο του Κιώτο και άλλες περιβαλλοντικές συμβάσεις καθορίζει την βάση για διμερή συνεργασία εδώ στη μετάβαση προς ε, μια οικονομία με χαμηλές εκπομπές του αερίου θερμοκηπίου και σε ε, οικονομίες που σέβονται το περιβάλλον και προσπαθούν να μειώσουν την, τα τη συνέψη αλλαγή του κλίματα, δημιουργούν το κατάλληλο πλαίσιο όπου μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτά τα θέματα και τα θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Βιετνάμ και αυτή η συμφωνία θα θέτει ένα νέο πλαίσιο για την προστασία των ευρωπαϊκών επενδύσεων στην, στο Βιετνάμ μαζί και το νέο σύστημα που έχουμε για το ε, αρμόδιο φορέα τη θέση διαφορών όσον αφορά τι επενδύσει. Προσβλέπω στι παρατηρήσει σα και ελπίζουμε να διατηρηθεί αυτή η ορμή για να συζητήσουμε περαιτέρω για το Βιετνάμ, για να κάνει το Βιετνάμ πολλέ μεταρρυθμίσει. Όσον αφορά τη ΣΥΠΑ τώρα, πριν από πέντε χρόνια περίπου, όταν ξεκίνησα τη θητεία μου, όλα τα θέματα τα εμπορικά αφορούσαν το TTIP, θα το θυμόσαστε κάποιοι από εσά. Αυτό υποτίθεται ότι θα ήταν ε, ε, ευρύτατη συμφωνία εμπορική μεταξύ Ευρωπαϊκής Ενώσεως και ΗΠΑ, ΕΕ που ήταν οι δύο μεγαλύτεροι εμπορικοί εταίροι. Ήταν δύσκολα τα πράγματα υπό την προηγούμενη Αμερικανική κυβέρνηση και κατέστη κάτι πολύ δύσκολο με τη νέα κυβέρνηση. Οι διαπραγματεύσει του TTIP έχουν κολλήσει και λόγω τη ανακοινώσεω των ΗΠΑ που θέλει να αποσυρθεί από τη Συμφωνία των Παρισίων, να αποσυρθούν οι ΗΠΑ, δεν βλέπουμε να υπάρχει κάποια δυνατότητα για μια πλήρη συμφωνία εμπορική με τη ΣΥΠΑ σήμερα και τα κράτη-μέλη στο Συμβούλιο επιβεβαίωσαν τον Απρίλιο όταν έδωσαν την εντολή για μικρότερη εμπορική συμφωνία επιβεβαίωσε ότι είναι απειρχιωμένη η εντολή και η συμφωνία, το, το TTIP. Όμω οι Ηνωμένε Πολιτείε είναι σημαντικός, ο σημαντικότερο εμπορικό μα εταίρο και εταίρο μα για τι επενδύσει και παρόλο που έχουμε εντάσει και δυσκολίε σε εμπορικέ μα σχέσει με αυτού, υπάρχει αμοιβαίο συμφέρον να διατηρηθεί ένα θετικό πρόγραμμα. Σχεδόν ακριβώ πριν από ένα χρόνο, ο πρόεδρο Γιούν και συνάντησε τον πρόεδρο Τραμπ στο Λευκό Οίκο για να συμφωνήσουν επί θετικού προγράμματο εργασιών και στα πλαίσια μια εκτελεστική ομάδα εργασία, όπω απεκλήθη. Υγήθηκα αυτή τη ομάδα πλευρά Ευρωπαϊκή και από τι πλευρά, είπα, πρέσβη Τάισερ, ε, ήθελε να ακολουθήσουμε διαφορετικά. Συμφωνήσαμε να ακολουθήσουμε πορείε, να μην έχουμε δασμού για βιομηχανικά προϊόντα, μικρότερη εμπορική συμφωνία, να προσπαθήσουμε να μειώσουμε τη γραφειοκρατία μέσω μια συμφωνία όσον αφορά την αξιολόγηση συμμόρφωση και ρυθμιστική συνεργασία επιθελοντική βάσεω σε διάφορου ε, τομεί. Επίση, αποφασίσαμε να κάνουμε μεταρρύθμιση του ΠΟΕ, να συνεργαστούμε πάνω σε αυτό, το κάνουμε αυτό μαζί με την Ιαπωνία και να προχωρήσουμε συγκεκριμένα χαρτοφυλάκια όπως σόγια, και φυσικό αέριο. Ε, αυτό εδώ και ένα χρόνο περίπου δημοσιεύουμε μία πλήρη έκθεση που θα δημοσιευτεί το τέλος αυτής της εβδομάδας και θα δημοσιοποιηθεί βεβαίως για να δώσουμε γενική εικόνα σχετικά με το που βρισκόμαστε όσον αφορά αυτά τα θέματα. Να σας πω πολύ σύντομα ότι όσον αφορά τη συμφωνία για τα βιομηχανικά αγαθά, ακόμα δεν έχουμε ξεκινήσει τι διαπραγματεύσει. η ΕΠΑ δεν είναι έτοιμε να ξεκινήσουν διαπραγματεύσει αν η Γεωργία δεν συμπεριληφθεί. Κάτι που είναι για μα κόκκινη γραμμή, οπότε για την ώρα τίποτα δεν συμβαίνει εκεί. Όμω για την εξολόγηση συμμόρφωση, όπου και το Συμβούλιο έδωσε εντολή τον περασμένο Απρίλιο πάνω σε αυτό, υπήρξαμε πιο καρποφόρε συζητήσει με τι ΗΠΑ για να διερευνήσουμε τη δυνατότητα οριζόντια συμφωνία που θα ήταν και για τι δύο πλευρέ. Συνομιλήσαμε οι συγκεκριμένου τομεί όπου θα μπορούσαμε να συνεργαστούμε χωρί να αλλάξουμε νομοθεσία ή κανόνε ή να μειώσουμε προδιαγραφέ. Σε τομεί όπω είναι οι ιατρικέ συσκευέ, η κυβερνοασφάλεια, φαρμακευτικά προϊόντα και συζητούμε σε εμπλεκομένου φορεί να εντοπίσουμε τομεί μελλοντική συνεργασία όπω εκτύπωση τριών διαστάσεων, ρομποτική κλπ. Κάποιοι τομεί Επίσης, συνεργαζόμαστε με τη ΣΥΠΑ και την Ιαπωνία για εξυγχρονισμό και επικαιροποίηση των κανόνων του ΠΟΕ, με άλλα λόγια, σε τομείς όπου ο ΠΟΕ δεν έχει κανόνες, να καλυφθούν κάποιες πολιτικές που ακολουθεί η Κίνα όσον αφορά τις βιομηχανικές ε, επιδοτήσεις και την υποχρεωτική διαβίβαση τεχνολογίας. Ε, έχουμε σημειώσει κάποια πρόοδο, αλλά δεν φτάσαμε στον επιθυμητό στόχο ακόμα σε αυτά. Ευπρόσδεκτη η απόφαση των ΗΠΑ να μην επιβάλλουν ακόμα τέλη σε αυτοκίνητα και ανταλλακτικά αυτοκινήτων, όμω η ίδια η έννοια ότι μπορούν να είναι θέμα απειλή τη εθνική ασφαλεία των ΗΠΑ, αυτό το επιχείρημα είναι παράλογο. Δεν θα δεχτούμε η αδίποτε διαχείριση του εμπορίου, ποσοστώσει ή εθελοντικού περιορισμού εξαγωγών. Και αν επιβληθούν οι δασμοί, εμείς θα έχουμε κατάλογο επανεξισορρόπησης που έχει προετοιμαστεί που έχει, αξίζει 35 δισεκατομμύρια ευρώ. Ελπίζω να μην χρειαστεί να το χρησιμοποιήσουμε αυτό το κατάλογο, όμως υπάρχει μια ιστορία παλιά με τα αεροσκάφη, μια σύγκρουση που χρονολογεί πριν από 15 χρόνια, μια μάχη μεταξύ Airbus και Boeing και ελπίζαμε αυτό το θέμα το ρυθμίσουμε στις σχέσεις μας και να ξεκινήσουμε την προσπάθεια εξέβρεση λύσεων. Τώρα που μιλάμε, η κυρία Βέιλαντ, η Γενική Διευθύντριά μου, είναι στη ΣΥΠΑ, ώστε να συζητήσουμε του ομολόγου του Αμερικανού, αν μπορούμε να βρούμε ένα αποτέλεσμα μέσω διαπραγματεύσεων του επόμενου μήνε. Αν αυτό δεν μπορέσει να γίνει, τότε οι ΗΠΑ θα επιβάλλουν δασμού σε εμά. Και πολύ σύντομα. Και εμεί σε αυτή περίπτωση, αλλά λίγο αργότερα θα ακολουθήσουν δικοί μα δασμοί για λόγου ιστορικού ε, ε, στην αντιμετώπιση αυτής της ιστορίας που είναι πολύ παλιά. Παρακολουθούμε τις σχέσεις από κοντά με τη ΣΥΠΑ. Και τέλος, Πρόεδρε, και εδώ καταλήγω, ε, το θέμα του ΠΟΕ, η κατάσταση στον ΠΟΕ είναι άκρως ανησυχητική. Έχουμε συνεχή απειλή μονομερών μέτρων που δεν είναι στα μέτρα του ΠΟΕ στα πλαίσια των εντάσσεων μεταξύ Κίνας και ΗΠΑ. Έχει μπλοκαριστεί ο διαρισμός των αρμοδίων για την επίλυση διαφορών στο όργανο έφεση από πλευρά ΣΥΠΑ και δεν μπορούμε να πάρουμε αποφάσει σε μεγάλο χρονικό διάστημα. Όπου ε, δεν είναι τέλειο. φορέας είναι το καλύτερο σύστημα που έχουμε. Χωρί αυτό θα επικρατούσε χάο. Γι' αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση με πολύ ισχυρή υποστήριξη από τα κράτη-μέλη και από το κοινοβούλιο σα και ήμασταν πολύ ενωμένοι σε αυτό, κινηθήκαμε για μια μεταρρύθμιση. Θέλουμε το φορέα έφεση να τον μεταρρυθμίσουμε χωρί να πειράζεται η κυριότητα αυτού και να υποβάλουμε μια πρόταση. Και όσον αφορά την καθημερινή εργασία του οργανισμού, αλλά και όσον αφορά, όπως ανέφερα, νέους κανόνες σχετικούς με τη δουλειά που κάνουμε με τη ΣΥΠΑ και την Ιαπωνία, αλλά και για την παρακολούθηση, κοινοποίηση, διαφάνεια κλπ. Εδώ συζητούμε με πολλά μέλη του ΠΟΕ και ελπίζουμε ότι τελικά θα καταλήξουμε σε κάποια θετική κατάληξη. Ε, ε περίπου με 80 χώρες έχουμε συζητήσει για διαπραγματεύσεις για την πολυμερή βάση για το ηλεκτρονικό εμπόριο, λίγο λιγότερα μέλη για τους εσωτερικούς κανονισμούς της υπηρεσίας, αλλά αυτό δείχνει ακόμα ότι ο ΠΟΕ είναι σε θέση να διαπραγματευτεί και να προωθεί διάφορα θέματα. Στόχος να ολοκληρωθεί συμφωνία όσον αφορά τις ελευτικές επιδοτήσεις στο τέλος του έτους, Δύσκολο αυτό αλλά εργαζόμαστε πραγματικά σκληρά πάνω σε αυτό το θέμα. Αυτά είναι τα θέματα τα οποία ήθελα να αναφέρω εν πρώτης, αλλά να γνωρίζω ότι υπάρχουν πάρα πολλά θέματα που αφορούν το εμπορικό θεματολόγιο και είμαι βέβαια στη διάθεσή σας για να απαντήσω ερωτήσεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ, εξότιμα μέλη και ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. The thing is that uh, we have now uh, seven speakers or seven coordinators on the list on behalf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 Μήπως μπορείτε να μας δώσετε περισσότερες ε, πληροφορίες σχετικά ε, με το θέμα αυτό και πώς είναι δυνατόν να ε, ενεργοποιηθεί ο μηχανισμός αυτός. Επίσης, η πρόεδρος Ούρσουνα Βόντεν Λάγεν αναφέρθηκε και στην συμφωνία. Έχετε κάποιες επιπλέον, επιπλέον στοιχεία ε, για να μας δώσετε σχετικά με την ε, ε, μεταδάση και σχετικά με την αποψήλωση. Ένα άλλο σημείο, θα είμαι σύντομος, για την Κίνα. Για την Κίνα γνωρίζουμε ότι υπάρχει το μεγάλο πρόβλημα της αφρικανικής επανόλης των χείρων. Δύο 200 εκατομμύρια ε, χείροι αναγκάστηκαν να ε, θανατωθούν. Αυτό όμως μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα ε, στους Ευρωπαίους παραγωγούς ε, όσον αφορά τώρα τον ΠΟΕ, αναφερθήκατε στα προβλήματα. Αυτό το δευτεροβάθμιο όργανο, ε, το όργανο ε, εφέσεων, ε, έχει μπλοκαριστεί. Ενδεχομένως γίνεται λόγος και για κάποιον ενδιάμεσο προσωρινό μηχανισμό. Έχετε να μας πείτε κάτι πάνω σε αυτό. Είναι σημαντικό να διατηρηθεί ε, αυτή η ορμή ε, ε, μεταρρυθμίσεων στον ΠΟΕ. Και πραγματικά τελευταία ερώτηση. Γνωρίζουμε ότι υπάρχουν ασάφειες όσον αφορά την υπόθεση Airbus Boeing. Πώς αντιμετωπίζετε αυτήν την ολοένα και κλιμακούμενη κατάσταση. Ευχαριστώ. 5,5 λεπτά αντί για 3. Εάν όλοι κάνουν το ίδιο πράγμα, τότε δεν θα έχουν οι τελευταίοι χρόνο να μιλήσουν. Ε, εξ των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πολλοί ζήτησαν το λόγο, όντως, αλλά αυτό σημαίνει ότι ε, τα επόμενα πέντε χρόνια τούτη η Επιτροπή θα είναι πάρα πολύ σημαντική. Εγώ θα προσπαθήσω να μην ξεπεράσω τα τρία χρόνια. Εγώ θα αναφερθώ κυρίως ε, στο Μερκοσούρ και άλλοι συνάδελφοι από την ομάδα μου θα αναφερθούν σε άλλα. Είναι πολύ σημαντικό θέμα αυτή η συμφωνία ε, Μερκοσούρ αλλά έχει αμφισβητηθεί και από πολλέ μη κυβερνητικέ οργανώσεις και από πολλού ε, εταίρου. Και εμείς λοιπόν ως ε, βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου οφείλουμε να συζητήσουμε κάποια θέματα. Ένα πολιτικό κύριο ζήτημα. Από τη μία μεριά ε, υπάρχει όντω πολύ καλή δουλειά στην Συμφωνία Μερκοσούρ, ας πούμε το θέμα του κλίματος, πάυση της αποψήλωσης, μείωση των εκπομπών, ε, συμφωνία των Παρισίων, κυρίως και όσον αφορά τη Βραζιλία όλα αυτά, αλλά από την άλλη μεριά υπάρχουν ζητήματα ε, που δεν είναι δυνατόν να τα ε, λησμονήσουμε και να αποστρέψουμε το βλέμμα μας. Πώς η Κομισιόν θα διασφαλίσει ότι η συμφωνία Μερκοσούρ θα ελέγχεται και πώς ε, θα ε, δεσμευθούν ε, οι εταίροι για τις υποχρεώσεις πρώτης επικύρωσης. Σημαντικό επίσης είναι το εξής, πώς μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι θα ενισχυθεί το κεφάλαιο TST. Και κάτι άλλο γιατί δεν είναι σαφές. Συμπεριλαμβάνεται και εξωτερική αναθεώρηση και έλεγχος από ε, εξωτερικούς ε, ανεξάρτητους ε, εμπειρογνώμονες και ποια είναι, ποιοι είναι οι μηχανισμοί, ποια είναι τα εργαλεία κυρώσεων που έχουμε στην διάθεσή μας και επίσης πώς και με ποιο τρόπο διαφοροποιείται το κεφάλαιο αυτό για το Μερκοσούρ σε σχέση με άλλες συμφωνίες. Επίσης, στην τεχνική ενημερωτική ε, συνάντηση με την τεχνική... Very last question on another... Ε, μας είχε γίνει αναφορά σε ένα ας πούμε κουμπί πανικού, ένα red ε, ε, button. Με ποιο τρόπο συγκεκριμένο μπορεί να υλοποιηθεί αυτό και επίσης θα, θα αφορά μονάχα θέματα διεθνούς εμπορίου ή θα αφορά και κάποιες παραβιάσεις οι οποίες μπορεί να γίνονται σε εσωτερικό επίπεδο. Και δεν αφήσα τελευταίο το θέμα της φορολόγησης και των φόρων. Πάρα πολύ ωραία. Τρία λεπτά μιλήσατε εξαιρετικά από την Renew Europe, Bro. Ευχαριστώ. Θα κάνω κάποιες γενικές παρατηρήσεις και μετά επιμέρους ερωτήσεις άλλοι συνάδελφοι της ομάδας. Γνωρίζουμε ότι η ευημερία, το εμπόριο οδηγεί ε, στην ευημερία. Οι πολίτες μας όμως ε, περιμένουν και κάποιες ε, εθνικές εμπορικές συμφωνίες και διεθνείς εμπορικές συμφωνίες να, και αναμένουν από αυτές να επιτύχουν και τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης. Πώς θα προχωρήσουμε έτσι ώστε καλύτερα να ληφθούν υπόψη αυτές οι προκλήσεις και στις τωρινές και στις μελλοντικές εμπορικές συμφωνίες. Οι διεθνείς εμπορικές οι συμφωνίες μπορούν να αποτελέσουν εργαλεία για τη βιώσιμη ανάπτυξη, εννοώ ε, και για τη, από οικονομική και οικολογική και κοινωνική ε, διάσταση και ταυτόχρονα να προωθούν την ανάπτυξη και την ευημερία Κατά την άποψή σας, πώς η συμφωνία Μερκοσούρ μπορεί να συμβάλλει ε, στην ανταπόκριση και σε αυτές τις ανάγκες και πώς μπορούμε να βοηθήσουμε τις χώρες αυτές. Δηλαδή, υπάρχει και η εναλλακτική να μην έχουμε ε, ε, συμφωνία και πρέπει να αναρωτηθούμε ε, είναι καλύτερο μήπως για τη βιώσιμη ανάπτυξη να μην έχουμε τέτοια συμφωνία. Επίσης, θα ήθελα την άποψή σας πάνω σε κάποια πρακτικά παραδείγματα, δηλαδή για τον τρόπο με τον οποίο οι εμπορικές συμφωνίες, ας πούμε Μερκοσούρα, αλλά και άλλες συμφωνίες με ποιο τρόπο οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και οι, ευρωπαϊκοί, οι ευρωπαίοι επιχειρηματίες μπορούν να ευεργετηθούν από αυτές τις συμφωνίες. Δηλαδή θα πρέπει να μετρήσουμε και πόσο αξίζουν αυτές οι συμφωνίες για την οικονομία μας, για τους επιχειρηματίες μας. Μπορείτε να μας δώσετε κάποια συγκεκριμένα στοιχεία, κάποια συγκεκριμένα αριθμητικά στοιχεία, κάποια συγκεκριμένα παραδείγματα έτσι ώστε ε, να αποτυπώσετε καλύτερα αυτά τα οποία σας ρωτώ. Ευχαριστώ. Thank uh, Εξ ονόματος των Πρασίνων, η κυρία Χαουτάλα. Ευχαριστώ, Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ε, νομίζω ότι εδώ θα πρέπει να βάλουμε και ένα πρόγραμμα τύπου ανταλλαγής εκπομπών, γιατί όταν μιλάνε πολύ οι πρώτοι δεν θα μείνει χρόνος για τους ε, δεύτερους. Εν πάση περιπτώσει, κυρία Επίτροπε, γνωρίζετε ότι εμείς εκτιμούμε ιδιαίτερα ε, τις ε, αρχές για το εμπόριο που φέρετε ήδη από το 2015. Φοβάμαι όμως ότι ε, ίσως θα πρέπει η επόμενη, ο διάδοχός σας ε, να έχει σαν μότο το Make Trade Not War, έτσι όπως εξελίσσονται ε, τα πράγματα. Είναι σημαντικό βέβαια η Ευρωπαϊκή Ένωση να υπεραμείνεται πάντα του ορθού εμπορίου και του ε, σωστού εμπορικού χώρου. Έχουμε δει τι σημαίνει Trade for All και είναι γεγονός ότι πρέπει να υπάρχουν οι απαραίτητες ε, δικλείδες ασφαλείας όσον αφορά την προστασία του περιβάλλοντος αλλά και το, την προστασία των εργαζομένων, προστασία των ε, δασών, την ε, ε, καταπολέμηση της παιδικής εργασίας ε, κλπ. Υπάρχουν πάντως κάποια ερωτήματα τα οποία προκύπτουν και νομίζω ότι θα πρέπει οπωσδήποτε να προχωρήσουμε στην υποχρεωτική, στις υποχρεωτικές δεσμευτικές έτσι ώστε να μπορέσουν όλοι ε, να ε, ευεργετηθούν από την ε, απόρρια αυτών των εμπορικών συμφωνιών και θα πρέπει οπωσδήποτε να υπάρξει μεγαλύτερη διαφάνεια, σεβασμός αξιών κτλ. Όσον αφορά τώρα τη συγκεκριμένη συμφωνία, να πω δύο λόγια για το Βιετνάμ. Εγώ ήμουν ε, εισηγήτρια για την FLECT που νομίζω ότι πραγματικά αποτελεί ένα πολύ σημαντικό εμπορικό εργαλείο και είναι καλό να το διευρύνουμε ακόμα περισσότερο. Χτες όμως πήρα μια απάντηση από τον πρόεδρο Τούσκ ε, σε ερώτησή μας ε, που αφορούσε ε, ζητήματα προστασίας ανθρωπίνων δικαιωμάτων στα πλαίσια της συμφωνίας με το Βιετνάμ. Θα επαναλάβω βέβαια ερωτήσεις που έχουμε ήδη υποβάλει. Πώς μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι οι βιετναμέζικες αρχές πριν από την από την σύμφωνη γνώμη του σώματος θα έχουν ήδη υλοποιήσει ε, όλα τα προαπαιτούμενα. Επίσης, ε, όσον αφορά το data localization, εάν υπάρχει πάντα αυτή η υποχρέωση, τότε οπωσδήποτε θα υποστούν κυρώσεις ε, οι επιχειρήσεις μας. Και κάτι τελευταίο για το Mercosur. Είναι 600 οι επιστήμονες και 300 οι ε, ηθαγενείς ε, οι οποίοι αναφέρονται ε, σε σεβασμό συγκεκριμένων δεσμεύσεων. Κάτι δεν πρέπει να μας πείτε και γι' αυτό. Από την ομάδα ID ο κύριος έχω κάποια ερώτηση πρώτα απ' όλα για τον παγκόσμιο ανταγωνισμό καθώς εδώ πέρα φαίνεται ότι παίρνουμε τον ρόλο αυτού ο οποίος ε, θεωρεί ότι έχει κάποια ηθική ανωτερότητα. Αυτό όμως σημαίνει μόνο ότι έχουμε κάποια ανταγωνιστικά μειονεκτήματα απέναντι παραδείγματος χάρη στην Κίνα. Πρώτα απ' όλα θεωρείται ότι η ισχυρότερη εστίαση αποκλειστικά στο εμπόριο και την οικονομία από χώρε όπως η Κίνα τις καθιστά πιο ελκυστικές από ό,τι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεύτερον, ποια μέτρα θέλετε να λάβετε συγκεκριμένα για να βελτιώσετε την ανταγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε παγκόσμιο επίπεδο για τις ε, επενδύσει. και για τα ζυζανιοκτώνα. Σε ποιο βαθμό γίνονται έλεγχοι και μπορούν να εμποδιστούν οι εισαγωγές προϊόντων που έχουν ψεκαστεί με ζανιοκτόνο που απαγορεύεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μπορείτε παραδείγματος χάρη να εγγυηθείτε ότι ο Ευρωπαίος καταναλωτής δεν θα καταλήγει να τρώει γλυφοσάτη από εισαγωγές. Και τέλος για τις μελλοντικέ ε, αποφάσεις. Θα ε, συνεχίσουμε να... Θα υπάρξει κάποιος μεγαλύτερος ρόλος συμβουλίου. ή θα συνεχίσουμε να έχουμε αυτή την κατεύθυνση της, ε, του παραγωνισμού των κρατών μελών. Ε, on e Σας ευχαριστώ από το ECR Μπουζόα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι. Βλέπουμε πως υπάρχει αυξανόμενος ε, προστατευτισμός, άρα έχει πολύ μεγάλη ε, σημασία το ελεύθερο εμπόριο για την ανάπτυξη, για τις ε, δουλειές. Εγώ είμαι από την ε, Φλάνδρα και μία στις τρεις θέσεις εργασίας ε, στη χώρα μας εξαρτάται από τις εξαγωγές. Συγκεκριμένα τώρα για τις ΙΠΑ έχω μία ερώτηση ελπίζω να υπάρξει κάποιο αποτέλεσμα και μία περιορισμένη έστω συμφωνία για τα βιομηχανικά αγαθά. Υπάρχει τουλάχιστον μια ελπίδα να συσταθεί το σώμα πρόσφυγων ε, του ΠΟΕ και να ληφθεί εκεί μια απόφαση για το Μερκοσούρ πάρα πολύ σημαντική η αγορά αυτή και συγχαρητήρια για την πρόοδο που επιτύχατε μετά από 20 ολόκληρα χρόνια και ελπίζουμε όπως και στην περίπτωση του Καναδά να έχουμε μία προώθηση, μία αύξηση της ανάπτυξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ανάπτυξης ε, και θέσεων εργασίας. Και κάτι το οποίο θα ήθελα να τονίσω σε σχέση με τον Brexit, ειδικά μιλάμε για σκληρό Brexit. Ελπίζω να έχουμε μία δυνατότητα για ευκολότερες ε, Ερώε και εξαγωγέ. Ειδικά στη Φιλάνδρα, αυτό αντικατοπτρίζει το εμπόριο δηλαδή με το Ηνωμένο Βασίλειο. Ένα 2,6% του ΑΕΠ μα τώρα. Υπάρχει φόβος για τις εισαγωγές κρέατος στην προκειμένη περίπτωση στη δικιά μας την χώρα όπου έχουμε και μία ποσόστοση για την ΣΕΤΑ έχουμε ένα 0,01% τη κατανάλωση κρέατος που εισάγεται. Τη ερώτησή μου λοιπόν είναι η εξής. Υπάρχουν κάποιες ε, προσδοκίες για μια περιορισμένη ποσόστοση του 1% η οποία δεν θα πληρωθεί. Και τελευταία ερώτηση για το χαρακτήρα αυτής της ε, συμφωνίας ε, σύνδεσης η οποία εξορισμού είναι κάπως περιορισμένη. Φοβάμαι ότι έτσι θα έχουμε κάποιες ε, δυσκολίες. Είχαμε και την απόφαση για τη Σιγκαπούρη όπου το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο είπε πως ε, θα πρέπει ε, να έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση αποκλειστική αρμοδιότητα για το διεθνές εμπόριο. Γιατί λοιπόν έχουμε αυτήν την περιορισμένη συμφωνία. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Και τώρα για την GUE ο κύριος Σόλτς. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και κάποιες ερωτήσεις ε, έχω να κάνω και εγώ, γιατί στο παρελθόν είχαμε εργαστεί έπαρκος για τα ζητήματα του δίκαιου εμπορίου και διαντολογικού εμπορίου. Και τώρα, μια που έχουμε συνάψει συμφωνία με Βιετνάμ και Μερκοσούρ, βλέπουμε πλέον ότι κορυφώνται αυτές οι προκλήσεις γιατί μιλάμε για παραγωγή, για εμπορικές σχέσεις μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτης χώρες και για κατανάλωση. Και αναφέρατε επίσης πως η συμφωνία του Μερκοσούρ ξεκίνησε πριν από 20 χρόνια και κανείς δεν, ε, εκτός από την λέσχη της Ρώμης ε, δεν μιλούσε τότε για κλιματική αλλαγή. Οπότε το ερώτημα είναι αν μπορούμε με το αποτέλεσμα αυτών των διαπραγματεύσεων να ανταποκριθούμε στις μελλοντικέ αυτές προκλήσεις, όχι μόνο την κλιματική αλλαγή, αλλά και στα αγαθά τα οποία θέλουμε να εμπορευτούμε. Ποιοι είναι οι όροι γι' αυτό. Αν μπορούμε να έχουμε τέτοια κατανάλωση στον 21ο αιώνα. Και έρχομαι στο ερώτημά μου στην συμφωνία της Μερκοσούρ έχετε δει την ατζέντα του 2030 του ΟΗΕ ως ένα μέτρο σύγκρισης. Κάποιες συγκεκριμένε ερωτήσεις τώρα. Πώς μπορείτε να διασφαλίσετε ότι η συμφωνία δεν θα παραβιάζει την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία για την ασφάλεια τροφίμων και ταυτόχρονα ότι ούτε η Βραζιλία ε, θα πρέπει να αλλάξει την εσωτερική της νομοθεσία. Αν και έχετε πει ότι υπάρχουν κάποια μέσα που περιέχονται στην συμφωνία. Μιλήσατε για χαμηλότερου δασμούς ε, ύψους 4 ε, δισεκατομμυρίων ευρώ του έτους, αλλά ταυτόχρονα θα μειώσουμε και εμείς τους δασμούς για την σόγια. Τι θα σημάνει αυτό λοιπόν για τους προπολογισμού των χώρων αυτών. Η Αργεντίνα, η Αργεντινή παραδείγματος χάρη, έχει ε, σχεδόν διπλασιάσει τις εξαγωγές της. Και τέλος για το Μερκοσούρι Για τις ε, συμβουλευτικές ομάδες εκεί της εγχώρης. θεωρείτε ότι οι εκπρόσωποι των αυτοχθόνων, των ΛΟΑΤΚΙ, των ανέργων εκπροσωπούνται και ότι είναι μια ανεξάρτητη διαδικασία για να αντιμετωπίσουν το αποτέλεσμα της εμπορικής συμφωνίας για τη δική τους πραγματικότητα. Πώς θα το διασφαλίσετε αυτό, ότι θα εργαστούν προς το συμφέρον μιας τέτοιας συμφωνίας. Ευχαριστώ πολύ. Τελευταίος, η κυρία Μπεγκίν. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και την Επίτροπο για την παρουσία της εδώ ε, σήμερα και την ευχαριστώ βέβαια και για τον τρόπο με τον οποίο διαρκώς ήταν ε, συμμετοχή στις εργασίες μας την προηγούμενη θα προσπαθήσω να είμαι ε, σύντομη, αλλά θα ήθελα να, σύντομη να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις για το Μερκοσούρ. Όσον αφορά γεωγραφικές ενδείξεις, ε, γιατί το κεφάλαιο για τη διανοητική ιδιοκτησία δεν έχει δημοσιευθεί με τα άλλα κεφάλαια και πότε θα δημοσιευθεί. Επίσης, έχουν λυθεί τα ζήτημα της μειομεγενούς εφαρμογής ε, της προστασίας γεωγραφικών ενδείξεων μεταξύ των διαφόρων χωρών. Δεύτερον, έχω την εντύπωση ότι λαμβάνοντας υπόψη ότι η διοίκηση Μπολσονάρο έχει ε, δώσει άδεια για την χρήση 150 ε, φυτοφαρμάκων ζεζανιοκτώνων. Ποιες ε, είναι οι προβλέψεις για την προστασία από τέτοιου είδους φυτοφάρμακα σε σχέση με τη διατροφική ασφάλεια. Τελε, μια τελευταία ερώτηση για το ρύζι. Σας ρωτώ λοιπόν ποιες είναι εάν υπάρχουν ε, ε, ε, σχέσεις όσον αφορά το ρύζι και την ρήτρα διασφάλισης για την Νοτιοανατολική Ασία. Επίσης, έχετε, έχετε κάνει εκτίμηση σχετικά με την γενική επίπτωση του Μερκοσούρ στον τομέα του ρυζιού. Τέλος, πώς είναι δυνατόν να ζητάμε ε, την ε, επαναχρήση, της, ε, επενεργοποίηση της ρήτρα πρόληψης όταν έχουμε περιπτώσεις όπως την αντίστοιχη ρήτρα, ας πούμε, για, για το ρύζι στη Συμφωνία με την Ανατολική Ασία. Επίσης, πάνω από ένα δίσε φαίνεται να έχουν προβλεφθεί έτσι ώστε να απαλληλθούν οι επιπτώσεις αυτής της συμφωνίας. Πρόεδρος, ε, προτείνω να δώσουμε στην Επίτροπο τον ε, λόγο για να απαντήσει μια, σε μια πρώτη φορά σε αυτές ε, τις ερωτήσεις. Βλέπω ότι πληθαίνει ο κατάλογος των ομιλητών. Δεν θα έχουμε χρόνο για όλους. Μια πρώτη φορά να απαντήσει η Επίτροπος και μετά συνεχίζουμε με το δεύτερο γύρο. Ευχαριστώ κυρίες και κύριοι βουλευτές. Θα προσπαθήσω να απαντήσω σε όλα. Πρώτα απ' όλα προς τον κύριο Χάνσεν για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις του Μερκοσούρ. Πράγματι υπάρχει ειδική παρόνοια για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Υπάρχει ειδικό κεφάλαιο σε όλες τις συμφωνίες που κάναμε που δεσμευόμαστε να τις διευκολύνουμε να υπάρχουν σημεία επαφής, ε, ε, site ε, κτλ. Για να διευκολύνουμε ακριβώ τη ραχοκοκαλιά της οικονομίας μας, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και Βεβαίως ε, θα πρέπει να είμαστε σε επαφή με τα επιμελητήρια, τις διάφορες επιτροπές για να διαχειριστούν αυτές οι πληροφορίες. Αυτό μπορούμε να κάνουμε. Για τις ε, δικλείδες ασφαλείας ε, όπως και σε άλλες συμφωνίες. Αν υπάρχει μια υπάρχει ακριβώς μια τέτοια ρήτρα. Όταν φτάσει στο ε, όριο αυτό σταματάει, δεν μπορεί να εξαχθεί περισσότερο. Ε, μπορούν οι αγρότες και οι λοιποί να λένε ότι υπάρχουν υπερβολικές εισαγωγές. Ε, σε αυτή την περίπτωση μπορούμε να κάνουμε κάτι. Υπάρχουν σχετικές διαδικασίες και θα δράσουμε. Βεβαίως υπάρχει ανάγκη για έρευνα για να φροντίσουμε ότι ε, θα δρούμε σύνομα, ε, εξάλλου πάντα το κάνει αυτό η Κομισιόν, αλλά μπορεί να ενεργοποιηθεί και από τις δύο πλευρές. Το κόκκινο αυτό κουμπί αφορά τις εισαγωγές. για την Κίνα και την Αφρικανική γρήπη των χείρων είναι μια καταστροφή αλλά μπορεί να σημαίνει ευκαιρίες για την Ευρώπη είμαστε σε επαφή με τις κινέζικες αρχές για να επιταχύνουμε την έγκριση των διαφόρων κρατών μελών για να υπάρξουν κάποιες δυνατότητες. Στην Γεωργία τελευταία έχουμε δει πως οι γεωργικές εξαγωγές έφτασαν το ύψος ρεκόρ των 12,8 δισεκατομμυρίων ευρώ πέρσι ε, και βεβαίως κύριοι στόχοι είναι Κίνα, ΗΠΑ, Καναδάς για την ενδιάμεση λύση για το Συμβούλιο Πρόσφυγής του ΠΟΕ. Αυτή τη στιγμή έχουμε το Γενικό Συμβούλιο στη Γενέβη του ΠΟΕ που συνεδριάζει. Ο πρέσβης Νέας Ζηλανδίας προσπαθεί να βρει κάποιον τρόπο να υπάρξει πρόοδος. Εάν αποτύχει αυτό θα μπορούσαμε διμερώς με τις ΙΠΑ να φτιάξουμε έναν προσωρινό μηχανισμό που θα έχει ακριβώς την ίδια μορφή με τους πόρους της γραμματείας του ΠΟΕ και θα επιλέξουμε ε, από τους ίδιους ανθρώπους ε, που ασχολούνται με την επιδιαιτησία ίσως συνταξιούχους δικαστές για να προστατευτούμε ακριβώς. Εν τω μεταξύ θα συνεχίσουμε να διασφαλίσουμε πως δεν θα σταματήσει να λειτουργεί τον Δεκέμβριο το εφετείο αυτό. και προσπαθούμε ακριβώ να έρθουμε σε επαφή με τη ΣΥΠΑ χωρί επιτυχία μέχρι στιγμή, ε, πρέπει να σα πω. Θα επανέλθω σε αυτό. Κυρία Φαν ρωτήσατε για τον φόρο στα σύνορα για τον άνθρακα στη χώρα μου. Ε, το έχουμε εδώ και δεκαετίες. Οπότε προσωπικά είμαι υπέρ αλλά εάν γίνει σε ευρωπαϊκό επίπεδο πρέπει να γίνει με τρόπο που δεν θα κάνει διακρίσεις. Είμαι υπέρ τη ιδέα, αλλά δεν θα το κάνει η δική μας επιτροπή, θα το κάνει η επόμενη, αλλά θα πρέπει να μην υπάρχει διακριτική μεταχείριση. Υπάρχουν θέματα ΠΟΕ. Αλλά νομίζω ότι η επόμενη επιτροπή μάλλον θα ξεκινήσει να εξετάζει το ζήτημα, ε, οπωσδήποτε συνεργασία και με από τη σκοπιά του εμπορίου, όπως σας είπα, θα πρέπει να μην υπάρχει διακριτική μεταχείριση. Για την αποδάσωση και τον Μερκοσουρή, η εμπορική συμφωνία από μόνη της δεν μπορεί να σύσει τον Αμαζόνιο βεβαίως. Δεν μπορούν να λυθούν όλα τα προβλήματα έτσι. Αλλά μπορεί να είναι ένα σημαντικό εργαλείο, γιατί στην εμπορική αυτή συμφωνία κάνουμε αναφορά σε όλα τα ζητήματα της Συμφωνίας των Παρισίων, της δεσμεύσεις της Βραζιλίας, στην απαγόρευση της αποδάσωσης, στην δέσμευση να ξαναφυτευτούν τα δάση και οι χώρες αυτές δεσμεύονται από τη Συμφωνία των Παρισίων και τις υπηρεσίες και επιπλέον είναι νομικά δεσμευτικό. Και μάλλον μέχρι το τέλος του έτους θα σας παρουσιάσουμε την αξιολόγηση μελέτη περιβαλλοντικού αντικτύπου της ε, συμφωνίας αυτής. Επίσης, έχουμε και νόμους στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την λαθροϊλοτομία. Ε, οπωσδήποτε θα το κοιτάξουμε και αυτό το θέμα. Πώς μπορεί τώρα να εφαρμοστεί. Επί χρόνια το συζητάμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυτό. Και δεν ε, στήριξε τις κυρώσεις η πλειοψηφία γιατί ακούγονται καλές κυρώσεις αλλά δύσκολα λειτουργούν στην πράξη και σε λίγες περιπτώσεις έχουν λειτουργήσει στην πράξη. Το μοντέλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι να είμαστε σε επαφή με την κοινωνία των πολιτών, με την κυβέρνηση. Να φτιάξουμε ένα πάνελ, κάτι το οποίο κάναμε τώρα με την Νότια Κορέα για τα εργασιακά. Το πάνελ θα συντάξει μια έκθεση δημόσια ε, κάτι το οποίο βεβαίως δεν είναι θετικό για την εν λόγω χώρα και για το επιχειρηματικό της κλίμα, για τη διεθνή της φήμη και ελπίζουμε έτσι να είναι εφαρμοστέα. Δεν μπορούμε να στείλουμε αστυνομία, αλλά υπάρχουν αυτά τα βήματα που σας είπα και βεβαίως θα υπάρχουν και πιο θετικές ε, πτυχές και νομίζω κάποιος το ανέφερε. Εάν κόψουμε τις επαφές με τις χώρες ε, θα είναι καλύτερο ή πως είναι καλύτερο να έχουμε ένα δεσμευτικό κείμενο και τις δεσμεύσεις των εταίρων μας π.χ. για το θέμα της διάσωσης του Αμαζονίου και τα ζητήματα αυτά. Γιατί κάποιες χώρες επιλέγουν το ένα, άλλες το άλλο. Εδώ πέρα τουλάχιστον τις δεσμεύουμε. Υπάρχει πάντα η πιθανότητα αναστολής της συμφωνίας. Μπορούν να το αποφασίσουν τα κράτη-μέλη αλλά υπάρχουν τρόποι να πιέσουμε. Νομίζουμε ότι θα λειτουργήσει αυτό στην περίπτωση της Νότιας Κορέας και ελπίζουμε και σε αυτή την περίπτωση. Οι εμπορικές συμφωνίες λοιπόν μπορούν να βοηθήσουν τα περιβαλλοντικά, τα εργασιακά. Βλέπουμε ότι οι χώρες κάνουν την προσπάθεια, αλλά βεβαίως δεν υπάρχει κάποια εγγύηση, δεν μπορούμε να αστυνομεύουμε άλλες χώρες. Οπότε είναι ένα σημαντικό εργαλείο σε συνδυασμό με τις άλλες χώρες, οικονομική διπλωματία και γιατί είμαστε σημαντική αγορά. Οπότε οι χώρες θέλουν να εμπορευτούν μαζί μας. Ε, ίσως ε, κάνουν πράγματα που δεν θα έκαναν με άλλες χώρες. Το έχουμε δει και με Καναδά, η Ιαπωνία. Έχει αυξηθεί τελευταία το εμπόριο, αλλά εντάξει είναι κάπως νωρίς για να δούμε ποιες θα είναι οι μεγάλες τάσεις για την Ιαπωνία. Δημιουργεί όμως θέσεις εργασίας, αυξάνει τις επενδύσεις και τις θέσεις εργασίας στην Ευρώπη. Για την δέουσα επιμέλεια γενικώ, ε, κυρία Χαουταλά, γνωρίζετε ότι η προσωπική μου προτίμηση είναι να κάνουμε περισσότερα, αλλά είναι περίπλοκο ζήτημα, πηγαίνει πέρα από το εμπόριο. Ελπίζω λοιπόν να θέσετε το ερώτημα αυτό σε μελλοντικού επιτρόπου ε, στου υποψηφίου. Για την κατάσταση ανθρωπίνων δικαιωμάτων με το Βιετνάμ, ναι, υπάρχουν σοβαρέ ανησυχίε για κάποια άτομα και για τον νόμο περί διαδικτύου. Το έθεσα στο Ανόη, στο υψηλότερο επίπεδο και η αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης θέλει ακριβώς να δει το νέο νόμο πριν εγκριθεί, οπότε κάνουμε ό,τι μπορούμε έτσι ώστε να υπάρχει ένας ε, ουσιαστικός διάλογος. Για τα ζανιοκτώνα, συγγνώμη, ήταν πολλές ερωτήσεις, ε, τα οποία είναι απαγορευμένα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα συνεχίσουν να παραμένουν απαγορευμένα. Πώς το ελέγχουμε. Ε, πρέπει να το ελέγχουν τα κράτη-μέλη και οι εταιρείε. Πρέπει να το κάνουν συνεχώ και πρέπει να υπάρχει εγγύηση ότι δεν θα χρησιμοποιούνται απαγορευμένα ζανιοκτώνα. Αν δεν μπορούν να το εγγυηθούν, μπορούμε να, ε, να τα απορρίψουμε στα σύνορα. Και αυτό συμβαίνει ήδη τώρα και δεν θα αλλάξει. Τα κράτη-μέλη είναι ενωμένα τελευταία στην εμπορική πολιτική. Όπως ε, ξέρετε, Είχαμε και την απόφαση του δικαστηρίου που είπε ότι για καθαρά εμπορικές ε, συμφωνίες ε, έχουμε ειδική πλειοψηφία κρατών μελών και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αλλά το κεφάλαιο για τις επενδύσεις πρέπει να εγκριθεί από όλα τα κοινοβούλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, η συμφωνία του Μαρκοσούρ είναι μια μεικτή συμφωνία, πρέπει να εγκριθεί από τα κράτη-μέλη, από εσάς και όλα τα εθνικά κοινοβούλια. Ελπίζω να εγκριθεί. Ναι, θα υποβληθεί. Για το Brexit δεν θα πω τίποτα. Μόλις ε, βγήκε καινούριος πρωθυπουργό στο Ηνωμένο Βασίλειο, θα περιμένουμε ε, κύριε Μπορζά να έρθουν προτάσεις από το Λονδίνο. Ας δούμε λοιπόν τι θα γίνει. Για το Μερκοσούρ απάντησα, είναι μια μεικτή συμφωνία. Η ποσόστοση για το κρέας είναι περιορισμένη και όπως σωστά είπατε έχει αποδειχτεί ότι οι Καναδοί έχουν χρησιμοποιήσει πολύ μικρό, ένα μισό της εκατό της ποσόστοσης γιατί δεν μπορούν να συμμορφωθούν με τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις ορμόνες παραδείγματος Οι ευρωπαϊκοί νόμοι ασφάλεια τροφίμων δεν θα αλλάξουν, κύριε Σούλτ. Και στην Αργεντινή και σε άλλες χώρες έχουν υπολογίσει ότι η εξαφάνιση των δασμών θα αντισταθμιστεί από τα ωφέλη του αυξημένου εμπορίου. Έχουν σίγουρα εξετάσει το θέμα σε εθνικό επίπεδο. Κυρία Μπεγκίν, για το θέμα της πνευματικής ιδιοκτησίας για το Μερκοσούρ δεν μπορώ να σας δώσω κάποια απάντηση. Είναι τεχνικά ζητήματα. Πρέπει να φροντίσουμε και οι τέσσερις χώρες να έχουν ακριβώς ε, τους ίδιους αριθμούς. Έχουμε εντατικές επαφές ε, και ελπίζω βεβαίως ακριβώς να ολοκληρώσουμε πριν το καλοκαίρι για τα ζανιοκτώνα το ίδιο. Για το ρύζι, όχι, κοιτάξτε, η Καμπότζη είναι κάτι τελείως άσχετο με το Μερκοσούρ ενεργοποιήθηκε το όριο αυτό μετά από πράγματα που μας είπαν οι καλλιεργητές ρυζιού της Ένωσης και ενεργοποιήθηκε αυτή η δικλίδα ασφαλείας. Δεν έχει δε μία σχέση όμως με το Μερκοσούρ. Uh, Ευχαριστώ. Μας μένουν 25 λεπτά περίπου και 15 ομιλητές. Ο καθένας από εσά πρέπει να τα καταφέρει σε 1,5 λεπτό. Αν τα καταφέρετε, η Επίτροπος έχει 2,5 λεπτά για να απαντήσει. Κύριε Γκέρι από το ΕΛΚ. Ευχαριστώ πολύ. Σχόλιο. Συγχαρητήρια όσον αφορά τη συμφωνία του το Βιετνάμ. Καλός λογικός συμβιβασμός. Δημιουργούνται ευκαιρίες στις μικρές επιχειρήσεις και μπορεί η βιομηχανία να παραμείνει στην Ευρώπη. Και για αυτούς που εξέφρασαν ανησυχίες τους συναδέλφους, Δεν θα λύσουμε όλα τα προβλήματα βέβαια, αλλά έχουμε πιθανότητες να έχουμε μια μόνιμη βάση διαλόγου με τις βιετναμικές αρχές. Ερώτηση για τη Συμφωνία Μερκοσούρ. Κάνουμε... Είμαστε στην αρχή της αξιολόγησης και κατανόησης της. Γεωργία. Τρία προϊόντα. Κοτόπουλο αποστομένο, βιοθανόλι, μέλι. Μας ανησυχούν όταν δημιουργηθεί το πλαίσιο υποστήριξης που ανέφερε και ο Επίτροπος Χόγκαν, ελπίζουμε ότι θα συμπεριληφθούν και οι γεωργοί που παράγουν αυτά τα προϊόντα για να μπορέσουν να ενταχθούν στο πλαίσιο υποστήριξης. Και αυτοί που θα είχαν υποστεί ζημιά από τη συμφωνία αυτή, οι γεωργοί, να πάρουν κάποια αποζημίωση, κάποια αντιστάθμιση των απολειών τους. Ευχαριστώ. Ο κ. Βάμπον. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ κυρία Επίτροπε, κυρία Μάνστρομ για τα όσα μας είπατε. Καταρχάς συγχαρητήρια. Ρηξικέλευτη η συμφωνία με το Μερκοσούρ. Οι εμπορικές σχέσεις μεταξύ Ευρωπαϊκής Ενώσεως και ΗΠΑ σε αυτή τη φάση είναι παράξενες. Οπότε αυτή η Συμφωνία Ελευθερών Συναλλαγών έχει μεγαλύτερη σημασία σαν η μεγαλύτερη εμπορική συμφωνία που έχει συνάψει ποτέ η Ευρωπαϊκή Ένωση, θα αυξήσει το εμπόριο και την ευημερία και στις δύο πλευρές, από τις δύο πλευρές του Ατλαντικού. Είμαι σίγουρος. Τώρα, πώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι συμφωνίες ελευθέρου εμπορίου προς όφελος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Υπάρχει δυνατότητα να χρησιμοποιηθούν οι κανόνες προέλευση τη συμφωνίας Ελευθέρου Εμπορίου προς διευκόλυνση τη κατάσταση για τι μικρομεσαίες επιχειρήσει. Ερώτηση. Τι κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να διευκολύνει τις μικρομεσαίες επιχείρησεις που χρησιμοποιούν αυτά τα μέτρα. Ευχαριστώ. Η κυρία Ρετζιμέντη έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ, κυρία Επίτροπε. Δράτω με τις, παρουσ... τις ευκαιρίες που είσαστε εδώ για να εκφράσω κάποιες σκέψεις γύρω από τη συμφωνία με το Μερκοσούρ και συγχαίρω τη Σάντρα Γκαλίνα, τη διαπραγματεύτρια από την Ιταλία για το επιτευχθέν αποτέλεσμα. Αυτή είναι ιδιαίτερα ευαίσθητη συμφωνία. Ε, τα μέτρα τα αμυντικά τα επιθετικά χρειάζονται πολύ λεπτή ισορροπία. Συγχαίρουμε για τη μείωση των δασμών και για το άνοιγμα κρισίμων τομέων, όπου εκεί είναι άριστα τα προϊόντα που φτιάχνονται στην Ιταλία. Ρύζι, ζάχαρη και κρέας είναι ε, προβληματική τομεί και έχει πληγεί η Ιταλία όσον αφορά αυτό. Μήπως πρέπει να γίνει ανάλυση αντικτύπου για κάθε χώρα τη Ευρωπαϊκή Ένωση, και ίσω και μία αξιολόγηση μετά, το περίοδο, μετά τον Brexit. Μπορεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εν σύντομα να έχει με τέτοια αξιολόγηση. Η συμφωνία θα καταφέρει να εφαρμόσει γρήγορα τα μέτρα, τα φυτογειονομικά και τους κανόνες προέλευσης. Συγκεκριμένο κίνδυνο είναι να υπάρχει σοβαρό αντίκτυπο για του καταναλωτέ τη Ευρώπη, Κάτι άλλο να διαδοθούν στην Ευρώπη νέα παράσιτα και ασθένειε που προέρχονται από τη Λατινική Αμερική είναι ένα κίνδυνο. Τέλο, ο Επίτροπο Χόγκαν αναφέρθηκε σε προληπτικά μέτρα για να μειωθεί ο αντίκτυπο ενδεχόμενο επιζήμια αποτελέσμα τη συμφωνία. Αναφέρθηκε σε ένα δισεκατομμύριο ευρώ. Μπορείτε αυτό να μα το διευκρινίσετε παραπέρα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Η κυρία Λαλίκ. Καλημέρα. Ευχαριστώ για τις απαντήσεις σας και την παρέμβαση. Είπατε ότι δεν είναι δυνατόν να έχουμε παντού αστυνόμευση για να εξακριβώνει ότι εφαρμόζονται κάποιες ρήτρε. Και έχετε δίκιο πάνω σε αυτό. Και είπατε ότι οι χώρες είναι έτοιμες να συμμετάσχουν και καταβάλουν προσπάθειες για τη σύναψη συμφωνίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί εμείς είμαστε μεγάλη αγορά. Να βάλουμε υπόψη δύο στοιχεία. Γιατί, εν τη αυτή περιπτώση, βασιζόμαστε να συνάψουμε κάποιες συμφωνίες και γιατί να μην πιέζουμε κάποιες χώρες όπως το Βιετνάμ, ούτω ώστε να δεσμευτούν πάνω σε θέματα κοινωνικά. Διότι πράγματι δεν μπορούμε να βάζουμε ένα αστυνομικό παντού σε αυτή τη χώρα εξακριβώνει ότι κάποιες ρήτρε γίνονται σεβαστές. Όσον αφορά το Βιετνάμ, γιατί να μην έχουμε απαιτήσει την απελευθέρωση κάποιων πολιτικών κρατουμένων. Γιατί να μην ζητήσουμε την κύρωση συμβάσεων πολύ βασικών του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας και να είναι πιο φιλελεύθερη η νομοθεσία. Έχουμε αρκετέ πιέσει που μπορούμε να ασκήσουμε. Είμαστε σημαντική αγορά. Και πάντα αναφερόμαστε στη σχέση μεταξύ αξία και διεθνού εμπορίου. Λέμε ότι μέσω του διεθνούς εμπορίου η Ευρώπη εξάγει τις αξίες τη. Εκεί θα ήταν σε ευκαιρία να το δείξουμε, κυρίω σπρώχνοντα προωθώντας το καθήκον ε, επαγρύπνησης περισσότερο. Πολύ γρήγορα, κατά την άποψή μου, αφήσατε εκτό αυτά τα θέματα. Και κάποιο συνάδελφο το ανέφερε αυτό να, πώς να φροντίσουμε να μπορέσουμε να πιέσουμε να υπάρχει επαγρύπνηση έναντι χωρών που είναι έτοιμε αρκετά εύκολα να διαπραγματεύονται μαζί μα, βλέποντα ότι έχουμε μεγάλο οικονομικό και πολιτικό κύρος και ισχύ. Ευχαριστώ. Ο κύριο Σούστα έχει το λόγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ κυρία Μάλμστρομ για αυτά τα οποία μας είπατε. Θα ήθελα να αναφερθώ στις συνομιλίες με τις ΙΠΑ. Πρώτα απ' όλα κάτι άλλο. Μέχρι τώρα απορούσα για το ότι είχε κάποιες απαιτήσει ο Γερμανός υπουργό Οικονομικών Altmaier, αλλά ε, δεν φανταζόμουν ότι θα ήθελα να αλλάξουν οι αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να κάνει τις αρμοδιότητες, να κάνουν τις αρμοδιότητες οι εθνικοί υπουργοί. να λίγο σοβαρά Ε, υπάρχει η δυσκολία του ότι οι ΙΠΑ δεν θέλουν να υπογράψουν την Συμφωνία των Παρισίων. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα υπάρχει καθόλου κεφάλαιο αηφορίας. Ακόμα και όταν μιλάμε για αγροποιημένο φυσικό αέριο, νομίζω ότι ακριβώ θα πρέπει να υπάρχει ένα τέτοιο κεφάλαιο. Δεύτερον, πώ έχουν τα πράγματα, γιατί μας, ε, από τη μία ο κύριο Γιούνκερ μα είπε ότι έχει ξεκινήσει η διαδικασία, αλλά μέχρι στιγμής δεν υπάρχει καμία διαπραγμάτευση επί της ουσίας των βιομηχανικών αγαθών, δηλαδή γιατί οι ΙΠΑ θέλουν να συμπεριλάβουν και τη γεωργικά προϊόντα. Και εμείς λέμε ότι δεν θέλουμε. Έχουν σταματήσει λοιπόν οι συνομιλίες. Τι σημαίνει αυτό. Έχει αποτύχει η στρατηγική. Γιατί από την άλλη ε, θέλαμε να παραμείνουν τα αυτοκίνητα εντός ε, και οι δασμοί τους οποίους εμείς θεωρούμε παράνομους ε, σε χάλιβα και αλουμίνιο ήθελαν ή ήπα να παραμείνουν. Όσον αφορά δε τη δική μας αντίδραση σε αυτούς τους ε, δασμούς ε, ποια είναι. Γιατί από ό,τι φαίνεται δεν προχωράνε τελικά καθόλου οι διαπραγματεύσεις. Ο κύριος Κέλλη. Ευχαριστώ πολύ τελευταία πέντε χρόνια έχω συμμετάσχει σε εργασίε τη Επιτροπή. Η Επίτροπο έκανε πολύ καλή δουλειά όσον αφορά τι εμπορικέ συμφωνίε. Είχα συμμετάσχει στι προσπάθειε τη συμφωνία με τη Σιγκαπούρη. Αυτά που λέει σήμερα είναι λογικά. Ένα τομέα με ανησυχεί ιδιαίτερα και του εκλογεί μου. Η συμφωνία Μερκοσούρ. Αχίλιο Πτέρνα είναι το περιβάλλον και η γεωργία. Είναι ηρωνικό το να ακούμε τα στοιχεία που γίνεται παράνομη υλοτομία στα τροπικά δάση και εμείς να διευκολύνουμε επιτρέποντας περαιτέρω είσοδο των χωρών αυτών στην ευρωπαϊκή αγορά. Όταν έχουν φτάσει στον πάτο οι τιμές του βοήου στην Ευρώπη, ε, μειώνεται η κατανάλωση και στη πατρίδα μου τα ζώα κατά κεφαλήν βγάζουν περίπου 200 ευρώ ή λιγότερο λόγω της μειώσεως κατανάλωσης και λόγω βεβαιότητος που σχετίζεται με τον Brexit. Από πλευράς γεωργικής, ο χρονισμός είναι ο χείριστος. Γι' αυτό αυτά πρέπει να τα λάβουμε υπόψη. Γιατί η διαδικασία κύρωσης. Αν κάθε κάτος μέλος πρέπει να κυρώσει, απαιτεί ομοφωνία. Και αν δεν κυρώσει ένα κάτος μέλος, θα σταματήσει τη συμφωνία. Αυτό σημαίνει. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο κ. Βατσικόφσκι. Το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ κυρία Επίτροπε, ευχαριστώ για την παρουσίασή σας. Ερώτηση για το Mercosur. Δύο ερωτήσεις. Μπερδεύτηκα. Μιλάμε για Συμφωνία Ελευθέρου Εμπορίου, μείωση δασμών. Ταυτόχρονα μιλάμε για ποσοστώσεις. Υπάρχουν ποσοστώσεις σε μια Συμφωνία Ελευθέρου Εμπορίου. Παράδοξο κατά την απόψή μου. Αν υπάρχουν ποσοστώσεις, μπορείτε να μου πείτε πώς θα διανεμηθούν στις χώρες αυτές οι ποσοστώσεις αυτός που έρχεται πρώτος παίρνει την ποσόστοση. Τι είναι, συμφωνία τύπου ντεόντα όπως έχουμε στο Κοινοβούλιο, πώς θα γίνει η κατανομή των ποσοστώσεων. Δεύτερο πρόβλημα. Σωστά καταλαβαίνω ότι παραδεχθήκατε ότι δεν έχουμε κανένα εργαλείο για να επιβάλλουμε τον σεβασμό των προδιαγραφών και προτύπων μας, των ευρωπαϊκών προτύπων και προδιαγραφών από τις χώρες αυτές. Μόνο μπορούμε να απευθύνουμε έκκληση και να δυσφημίσουμε την Βραζιλία στην Ευρώπη, καταστρέψουμε τη φήμη της, προβάλλοντας κάποια κακή τη συμπεριφορά αν αυτή λάβει χώρα. Σας ευχαριστώ. Η κυρία Μακουλάτα. Ευχαριστώ πάρα πολύ ε, κύριε Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, ευχαριστούμε που είστε εδώ μαζί μας. Τρεις ερωτήσεις ε, για το Μερκοσούρ, για τον ΠΟΕ και για τις Ηνωμένε Πολιτείε. Ε, όσον αφορά το Μερκασούρ, συγχαρητήρια γιατί ξεκίνησε μια συμφωνία η οποία γεωπολιτικά και στρατηγικά είναι πάρα πολύ σημαντική και παίζει μεγάλο ρόλο άλλωστε και στην εμβάθυνση του ρόλου της Ευρωπαϊκής Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Λατινική Αμερική. Όσον αφορά τη βιώσιμη ανάπτυξη όμως, δεν κατάλαβα πολύ καλά σε περίπτωση που ε, οι δεσμευτικά υποχρεωτικές ε, ε, προβλέψεις, οι πρόνοιες δεν γίνουν σεβαστές. Τι θα συμβεί εάν δηλαδή πώς θα λειτουργήσει κατά την έννοια αυτή ε, ο μηχανισμός επίλυσης ε, συγκρούσεων και προβλημάτων. Δεν το κατάλαβα πολύ καλά. Ένα άλλο θέμα το οποίο έχει γίνει καλά είναι ε, αυτά τα δελτία τα οποία μπορούν να διευκολύνουν την κατανόηση θεμάτων Εβραίων. Αλλά δεν το είδα όμως στη συμφωνία. Σε ένα δελτίο αναφέρεται στην ανάγκη συνεργασίας έτσι ώστε το ε, εμπόριο να υποστηρίξει ε, τις ε, αλυσίδες προμήθειας κατά της αποψήλωσης. Αυτό από πλευρά εμπορική πώς θα το λύσετε, δηλαδή πώς θα γίνει πραγματικά. Επίσης, όσον αφορά την συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών στους μηχανισμούς παρακολούθησης της συμφωνίας. Πώς ε, θα το σχεδιάσετε αυτό, πώς θα το καθορίσετε. Ε, είχα την ευκαιρία να μιλήσω με εκπροσώπους ε, κοινωνίας των πολιτών και με συνδικάτα στις χώρες αυτές και διαπιστώνω ότι έχουν αρκετά επικριτική στάση όσον αφορά τον μηχανισμό. Γι' αυτό λοιπόν δεν ξέρω έχετε κατά νου τις επικρίσεις αυτών των εκπροσώπων. Φαντάζομαι ότι φτάσανε στα αυτιά σας. Όσον αφορά την ε, ε, γεωργία, υπάρχουν γεωργικοί τομείς που δεν θεωρούνται ευαίσθητοι, αλλά που πιστεύω ότι αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα περίπλοκη κατάσταση. Ε, αναφέρομαι κυρίως στα σπεριδοειδή, τα οποία έχουν ε, υποστεί πολύ μεγάλη κρίση, λαμβάνοντας υπόψη και την ε, τη γενική διεθνή κατάσταση. Είναι γεγονός πάντως ότι ε, η κατάσταση δεν είναι ίδια με τρία χρόνια πριν. Ε, δεν ξέρω εάν θα ληφθεί υπόψη ε, και ε, ο συσσωρευμένος αντίκτυπος ε, και επίσης πώς θα εφαρμόσετε τη Συμφωνία Μερκοσούρ σε ένα ήδη προβληματικό τομέα, αλλά δώσει υπόψη και τη μελέτη αντικτύπου που θα δημοσιευθεί το φθινόπωρο. Ε, επίσης, ε, ε, κάποιες, κάποιοι μηχανισμοί που προληπτικά θα μπορούσαν να λειτουργήσουν πριν υπάρξει ζημία η Κομισιόν μπορεί να ξεκινήσει τις διαδικασίες αυτής. Εμείς έχουμε πει ότι ε, δεν θα πρέπει μονάχα ο τομέας να έχει το βάρος της ε, απόδειξης. Θα μπορούσε να γίνει κάτι αντίστοιχο και στην προκείμενη περίπτωση. Ε, εάν, ας πούμε, δούμε ότι έχουμε πολύ ψηλότερες εισαγωγές από αυτές που θα είχαμε ε, προβλέψει με ποιο τρόπο ε, το κόστος θα μπορούσε να, ε, και η επίπτωση θα μπορούσε να μειωθεί. Σε περίπτωση παραβίασης των φυτογειονομικών όρων, η μόνη λύση σε περίπτωση που δεν υπάρχει συμμόρφωση με τους ευρωπαϊκούς κανόνες είναι να σταματήσει η εισαγωγή ή θα εφαρμοστούν προληπτικά μέτρα. Τέλος, όσον αφορά τον ΠΟΕ. Μπορείτε να μας πείτε δύο λόγια παραπάνω σε περίπτωση που δεν καλυφθούν οι θέσεις, δεν διοριστούν δηλαδή οι δικαστές, υπάρχουν ε, εναλλακτικές λύσεις όσον αφορά την επίλυση των διαφωνιών. Ευχαριστώ κύριο Μόργαν Σάντσες και έχω την κυρία Άντερς, τον κύριο Καβατσίνη, τον κύριο Βίτρια, τον κύριο Κάγιας, τον κύριο, την κυρία Ραφαέλα και τον κύριο Μπουτικόφερ. Κύριε Μόργαν Σάντσες. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Καλώς ορίσατε κυρία Επίτροπε. Ε, είναι πραγματικά επιστροφή στο μέλλον. Ήμουν πριν από 10 χρόνια σε αυτήν την επιτροπή και βλέπω ότι εδώ και 10 χρόνια δεν έχουν αλλάξει ορισμένα πολύ καυτά θέματα. Όσον αφορά το Μερκοσούρ, υπάρχουν δύο πυλώνες, ε, πολιτικοθεσμικός και ε, συνεργασίας. Ε, είναι καλό να αρχίσει να ισχύει μάλιστα αυτό όσο γίνεται περισσότερο, γιατί έχουμε ανθρώπινα δικαιώματα, κλίμα και λοιπά Θέματα πάρα πολύ σημαντικά. Η κλιματική αλλαγή είναι σημαντική, πρέπει να προχωρήσουμε. Έχετε κάποιο χρονοδιάγραμμα επικύρωσης από πλευρά των κρατών όσον αφορά το θέμα αυτό. Δεύτερη ερώτηση. Σε σχέση με τις Ηνωμένε Πολιτείες και την Κούβα. Υπάρχει ε, μία ε, διαφωνία που από το 90 ε, είχε αποσιωπηθεί κατά κάποιο τρόπο, αλλά αυτή το δόγμα Χένς Μπόρτον έχει αναζωοποιηθεί και αναβιώσει από τον πρόεδρο Τραμπ. Έχετε κάποια λύση όσον αφορά το θέμα αυτό, γιατί ασκούνται πράξεις οι οποίες είναι κατάφορα παραβιάζουν την διεθνή νομιμότητα. Ευχαριστώ η κυρία Άντερσον. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Πρέπει να σας πω ότι αυτή η προσέγγιση σας, σας περιμένουμε να δούμε για τον Μπόρις Τζόνσον, δεν ε, ικανοποιεί τους εμπορευόμενους, κυρίως στην Ιρλανδία, τη Βόρεια Ιρλανδία. Ε, προβληματίζονται γιατί ο Μπόρις Τζόνσον φοβούνται ότι θα υλοποιήσει τις προεκλογικές του θέσεις ε, και επομένως θα αντιταχθεί στην ε, βούληση των πολιτών έτσι όπως ελεύθερα εκφράστηκε. Ε, όσον αφορά τις ε, συμφωνίες, ε, την συμφωνία αυτή, πιστεύετε ότι υπάρχει οποιαδήποτε ελπίδα ότι θα αποσοβηθεί το ενδεχόμενο του σκληρού Brexit και του σκληρού συνόρου στην ε, Ιρλανδία γιατί αυτό προβληματίζει ε, πάρα πολύ λαμβάνοντας υπόψη ότι ε, υπάρχουν οι συμφωνίες της Μεγάλης Παρασκευής, τις δημοκρατικά αποδεκτές συμφωνίες και επομένως θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει πιστεύουμε ότι και η Επιτροπή μας εδώ αλλά και άλλες επιτροπές ε, θα πρέπει να το μελετήσουν το θέμα αυτό και το οφείλουν ε, και στου στον λαό της, ε, στους πολίτες της Ιρλανδίας όσον αφορά το θέμα των κυρώσεων ε, σε περίπτωση ε, παραβιάσεων σε σχέση με τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης. Είπατε προηγουμένως ε, ότι το Συμβούλιο παρενέβη εναντίον αυτής της αρχής. Θα πρέπει να, τα ξέρουμε τα θέματα αυτά. Ευχαριστώ πολύ και θέμα διαφάνειας των διαδικασιών. Ευχαριστώ κυρία Καβατσίνη. Σα ευχαριστώ κύριε Επίτροπε, ευχαριστώ και τους συναδέλφους για τις ενδιαφέρουσες ερωτήσεις. Συμφωνώ μαζί σας όταν λέτε ότι οι εμπορικέ συμφωνίες δεν μπορούν να λύσουν όλα τα προβλήματα του κόσμου, σωστό. Αλλά θα μπορούσαμε να είμαστε κάπως πιο φιλόδοξοι. Όπως είπε η συνάδελφος πριν, οι περισσότεροι από τους εταίρους θέλουν να εμπορευτούν μαζί μας και έχουμε αυτό το τεράστιο πλεονέκτημα. Και ε, νομίζω ότι θα έπρεπε να είμαστε κάπως πιο φιλοδοξοί. Είπατε και η κυρία Καλίνα είπε παραδείγματος χάρη Μερκοσούρ, ε, Συμφωνία των Παρισίων ε, και η αρχή της προφύλαξης έχουν ενταχθεί στην συμφωνία. Όταν μιλάμε όμως με Βραζιλιάνους μας λένε ότι ναι, έχουμε περιορίσει αυτές τις αρχές στις διαπραγματεύσεις. Μήπως λοιπόν δεν έχετε καταλάβει το ίδιο πράγμα οι δύο πλευρές και εάν σας κατάλαβα σωστά είπατε παραδείγματο χάρη αν χρησιμοποιηθούν ζυζανιοκτώνα στην Βραζιλία σε κάποια προϊόντα είμαστε 100% σίγουροι ότι θα σταματήσουν στα σύνορα και δεν μπορούν να εισαχθούν. Ε, ισχύει αυτό και για προϊόντα τα οποία προφανώς έρχονται από αποδασωμένες περιοχές γιατί η υπουργό μου από την Γερμανία είπε ότι για τη σόγια ότι δεν θα ε, εισάγουμε σόγια στην Ευρωπαϊκή Ένωση ε, που έχει φυτευτεί σε αποδασωμένη περιοχή. ισχύει αυτό. Και τέλος, σύμφωνα με τις δικές μας προβολές, ε, η παραγωγή βοήου κρέατος ή αυτοκινήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα αυξηθεί, γιατί θα έχουμε περισσότερες εξαγωγές αυτών των προϊόντων. Πώς συμβιβάζεται αυτό με τους στόχους ε, για τους οποίους έχουμε δεσμευτεί στην Συμφωνία των Παρισίων. Είναι κλάδι έντασης διοξιδίου του άνθρακα. Εάν αυξηθεί η παραγωγή βοήου κρέατος, παράγουμε περισσότερο διοξιδίου του άνθρακα. Πώς συμβιβάζεται αυτό με τις συμφωνίες ε, τις οποίες έχουμε υπογράψει. Ο κύριος Βίνκλερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε. Πρώτα απ' όλα να σας συγχαρώ για τη δουλειά που κάνετε και να συγχαρώ και τις υπηρεσίες σας για την δουλειά που έκαναν. Πολύ σημαντική. Έχουν επιτύχει σημαντικά αποτελέσματα για τα κράτη-μέλη, για τις εταιρείες, για τους πολίτες μας, για τις δουλειές, για τους νέους κτλ. κτλ. Να ρωτήσω και κάτι άλλο, γιατί πρέπει από μετά από πέντε χρόνια βέβαια η εντολή σας λίγη και η στρατηγική εμπορίου για όλους ε, επίσης ε, θα ε, κάνετε κάποια έκθεση εφαρμογής, κάποια αξιολόγηση γιατί η προσωπική μου άποψη είναι και νομίζω η πλειοψηφία του ΕΛΚΟ ότι ήταν μια καλή στρατηγική ήταν η κατάλληλη στρατηγική για το ευρωπαϊκό συμφέρον αλλά να δούμε όλοι αν ισχύει αυτό πράγματι μετά για την επιβολή. Και αυτό είναι μια συζήτηση που θα συνεχιστεί στην Επιτροπή μας. Και βεβαίως εγώ ανήκω σε αυτούς ε, που θεωρούν ότι η εφαρμογή των ρητρών βιωσιμότητας ε, ε, μπορεί να γίνει μέσω του μέσου συνεργασίας αλλά μπορείτε να ζητήσετε από τις υπηρεσίες σας να δημοσιεύσουν και κάποια στοιχεία για τα μέσα εμπλοκής με τους εταίρους στην βιομηχανία μας κτλ. και στην κοινωνία των πολιτών και τα σχετικά. Και δύο σύντομε ερωτήσεις. Έχετε κάποιο χρονοδιάγραμμα ή κάτι το οποίο θα θέλατε για τη σχέση με το Βιετνάμ, ε, οι υπηρεσίε σας ε, έχουν κάνει κάποιες σκέψη. και τέλο. η Κίνα. Νομίζω μιλήσαμε λίγο για την Κίνα. Η Κίνα βέβαια απασχολεί κάθε συζήτησή μας γιατί είναι πάρα πολύ σημαντική. Θεωρώ λοιπόν ότι τον Μάρτιο εμείς ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρούμε την Κίνα έναν συστημικό αντίπαλο Είδατε λοιπόν κάποια αλλαγή στην συμπεριφορά των Κινέζων εταίρων και θα μπορούσαμε να ελπίζουμε ε, σε κάτι στο επόμενο έτος. Φέτος μάλλον όχι, αλλά του χρόνου κάποιες διαπραγματεύσεις ή τουλάχιστον κάτι για τις γεωγραφικές ενδείξεις που μας υποσχέθηκαν. Σας ευχαριστώ. Σχεδόν τελειώσαμε οι τρεις τελευταίοι ομιλητές και ως κανιάς. χωρίς μικρόφωνο. Intentaré ceñirme yo sí al minuto 30. Ναι, και εγώ 3,5 λεπτά θα μιλήσω. Πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω την Επίτροπο για την ε, ηγετική της συμπεριφορά, τα πολύ καλά αποτελέσματα, την ε, σοβαρή της δουλειά. Νομίζω πρέπει να τα αναγνωρίσουμε αυτά ε, σε μια ιδιαίτερη στιγμή πολύ σημαντική για την ηγεσία αλλά και για την ηγετική θέση της Στρατηγικής Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή βρισκόμαστε σε μια

Ε, Μερκοσούρ ε, ε, σχετίζεται και με τα προβλήματα τα οποία έχουν συνήθως αυτού του είδους οι μεγάλες συμφωνίες. Δηλαδή αυτού του είδους οι συμφωνίες πολλές φορές υποδαβλίζουν φόβους, συζητήσεις για προστατευτισμούς, φόβους λοιπόν που αναβιώνουν ας πούμε στο πνεύμα των πολιτών και που εν τέλει αποδεικνύουν και ότι λείπουν πολλές φορές κάποιες σωστές ρήτρε, ε, ας πούμε το θέμα των εσπεριδοειδών ή κάποιες προστασίες για συγκεκριμένα πράγματα. Ε, ε, κάποιες, ας πούμε το θέμα των εσπεριδοειδών είναι γεγονός ότι εδώ έχουμε πτώση 25% των τιμών. Είχαμε επίσης και τη φαιά κοιλίδα η οποία δημιούργησε ακόμα μεγαλύτερα προβλήματα. Είναι γεγονός ότι μπορούν να βελτιωθούν και η διαφάνεια των μηχανισμών, αλλά θα πρέπει να δούμε και πώς μπορούμε να βελτιώσουμε και τους μηχανισμούς ε, ε, για τις ρήτρες ε, προστασίας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, κυρία Επίτροπε. Είπατε ότι χωρίς τον ΠΟΕ θα επικρατούσε χάος στο εμπόριο. Αν δεν μπορείτε να καταλήξετε θετική συμφωνία με τις ΗΠΑ για πολυμερές εμπόριο, πώς μπορείτε να υπερασπιστείτε τη θέση μας έναντι των πράξεων της Αμερικανικής κυβερνήσεως. Μια συμφωνία με τις χώρες Μερκοσούρ έχει αντίκτυπο όσον αφορά τις υπερπόντιες, ε, τα υπερπόντια εδάφη και επικράτειες. Δεν ξέρω ακόμα τι είδους αντίκτυπο. Από ό,τι ξέρω, οι Ολλανδικές υπερπόντιες εκτίσεις δεν έχουν ενημερωθεί όσον αφορά τις διαπραγματεύσεις, κατά τη διάρκεια διαπραγματεύσεων. Μπορείτε να εγγυηθείτε, είστε πρόθυμοι να κάνετε συγκεκριμένη εξολόγηση αντικτύπου για αυτή την περιοχή ε, σε συνάρτηση με τη Συμφωνία Μερκοσούρ. Ευχαριστώ κ. Μπιτικόφερ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Um, Επίτροπε Μάλστρομ, να θέξω και εγώ για, την ομασία προέλευσης και την Κίνα. Θα μπορέσουμε να συνάψουμε πριν το τέλος του έτου συμφωνία. Αυτή είναι η πρώτη ερώτηση. Δεύτερη. Στην κυβέρνηση Τραμπ, όλο και οι περισσότερες φωνές ζητούν αποσύνδεση από την Κίνα. Οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις κινδυνεύουν να πέσουν θύμα αυτής στρατηγικής αποσύνδεσης. Έχετε κάποια στατηγική να το αντισταθμίσετε αυτό. Τρίτη ερώτηση. Όσον αφορά τη γενική θέση των είπα ότι ποτέ δεν θα συνάψουν συμφωνία για βιομηχανικά αγαθά χωρίς να συμπεριλάβουν κάποια άλλα στοιχεία, πώς μπορεί να γίνει η διαπραγμάτευση. Thank Uh, Ευχαριστώ. Και εγώ έχω μια ερώτηση, αλλά ο κύριος Βίνκλερ την έθεσε α, θεμού. Είναι η Συμφωνία Ελευθέρου Εμπορίου με το Βιετνάμ η ερώτησή μου. Το χρονοδιάγραμμα αυτή ήταν η ερώτησή μου. Αν μπορείτε να απαντήσετε παρακαλώ κυρία Επίτροπε. sorry. Ναι, συγγνώμη. Κοίταγα τις σημειώσεις μου. Κύριε Κέρι, για την ερώτησή σας ε, για το Σύριο Σκοτοπουλού έχουμε 800.000 τόνους πλεόνασμα εξαγωγών. Τώρα το λίγο που αφορά το Μερκοσούρ δεν είναι πρόβλημα. Για το μέλι εισάγουμε ακόμα το 45% των όσων καταναλώνουμε. Σύμφωνα με κάποιους πρώτους υπολογισμούς, οι εισαγωγές από το Μερκοσούρ θα αντικαταστήσουν αυτές ε, της Κίνας. Οπότε δεν θα μας επηρεάσει. Και γιατί είναι εθανόλη, είναι βιομηχανική εθανόλη που χρειαζόμαστε. για το δίκτυο στήριξης ε, του κυρίου Φιλχόγκαν ε, νομίζω είναι σε μια διπλανή αίθουσα. Ε, δεν το γνωρίζω, αλλά τα επεξεργάζεται οπωσδήποτε η Κομισιόν και θα σας παρουσιαστούν μόλις είναι έτοιμα. Για τους κανόνες προέλευσης. Ναι, στις περισσότερες περιπτώσεις με το Μερκοσούρ οι κανόνες είναι οι ευρωπαϊκοί. αυτό διευκολύνει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις μας και ακριβώ προσπαθούμε να βασιστούμε στην ευρωπαϊκή προσέγγιση. Γιατί είναι βασικό αυτό για τις μικρές εταιρείε ε, για να μην έχουν δύο γραμμές παραγωγής. Για το θέμα του Brexit ε, δεν θα απαντήσω, πρέπει να ξεκαθαρίσει ακόμα το θέμα, το τι θα γίνει, τι θα πει ο νέος Πρωθυπουργός, τον κύριο Μπαρνιέ. Είμαι σίγουρος ότι ο κύριος Μπαρνιέ ευχαριστώ θα έρθει στην Επιτροπή σας, ε, το κάνει πάντα πρόθυμα θα απαντήσει σε μερικές εβδομάδες. Ε, κυρία Λουλή, για το Βιετνάμ. Η πρώτη σύμβαση που εδώ και μερικές εβδομάδες υπεγράφει από το Βιετνάμ χάρη στην πίεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι υπόλοιπε που απομένουν έχουμε δέσμευση γραπτή από την κυβέρνηση με προθεσμία το 2021 και το 2022 νομίζω, σε μια επιστολή αναφέρεται που διαβίβασα στην Επιτροπή σας και πιστεύω ότι χωρίς την πίεση που ασκήσαμε κατά διάρκεια των διαπραγματεύσεων και για τη διαδικασία της επικύρωσης αυτό δεν θα είχε γίνει όσον αφορά τον νόμο των άλλων για, για, τα, για τον κυβερνοχώρο. Έχουμε έρθει σε επαφή με την κυβέρνηση και τα Υπουργεία στο Βιετνάμ για αυτό το θέμα και η αντιπροσωπεία μα στο ΑΝΟΙ καταβάλει προσπάθειες για να γίνουν ιδέωσες τροπολογίες όσον αφορά την νομοθεσία που για μας δημιουργεί πολλά προβλήματα και ερωτηματικά. Και όσον αφορά κάποια ανθρωπιστικά ζητήματα, και εκεί εγώ και ο κύριος Γιούνκερ και ο κύριος Τούσκ θέσαμε αυτά τα θέματα επανειλημμένα, προσπαθούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτό το παράθυρο που έχουμε, αυτό το άνοιγμα που έχουμε αυτή τη στιγμή, για να πιέσουμε την κυβέρνηση του Βιετνάμ για την ενδιάμεση λύση του ΠΟΕ. Δεν υπάρχει κάποιο σχέδιο Β που μπορούμε να έχουμε έτοιμο γιατί το εφετείο τρόπο βασίζεται ακριβώς στο ότι υπάρχει ένας δεύτερος βαθμός προσφυγής και αυτό έχει λειτουργήσει με τις περισσότερες χώρες του ΠΟΕ. Τώρα, θα σταματήσει όμως να λειτουργεί στις 12 Δεκεμβρίου αν δεν συμβεί τίποτα. Αυτό είναι ατυχέστατο. Και συνεχίζουμε να κάνουμε επαφές διμερείς ε, και με τη ΣΥΠΑ για να ξεμπλοκαριστεί ακριβώς ο διορισμός των επιδιωτητών αναγνωρίζοντας ότι μπορεί να επέλθουν κάποιες βελτιώσεις ε, χωρίς να αμφισβητούμε την ακαιρεότητα του συστήματος των δύο επιπέδων. Μέχρι στιγμής δεν έχει αλλάξει τίποτα. Γι' αυτό αρκετές χώρε αποφάσισαν να πούν μήπως να φτιάξουμε κάτι ε, παράλληλο σαν και αυτό στην περίπτωση που συγκρουστούν οι δύο πλευρές. Μπορούμε να το κάνουμε, αλλά πρέπει να υπάρχει μια κρίσιμη μάζα χωρών, κάτι το οποίο σήμερα δεν φαίνεται να υπάρχει. Οπότε μπορούμε να συνεργαστούμε με κάποιες ε, χώρες κλειδιά, κάτι το οποίο θα είναι μια ενδιαφέρουσα ενδιάμεση λύση. Άλλες χώρες διμερώς μεταξύ τους έχουν αποφασίσει να μην ζητήσουν ποτέ μια δεύτερη γνώμη. Αυτό είναι κακή ιδέα. Χρειαζόμαστε δύο επίπεδα, νομίζω. Γι' αυτό ακριβώς συζητάμε με τον Καναδά και με άλλους εάν αυτό θα μπορούσε να αποτελέσει μια λύση. Για την κύρωση της Συμφωνίας Σύνδεσης, κύριε Μορένο. Κανονικά τίθεται ενισχύει ταυτόχρονα με τη Συμφωνία Ελευθερίου Εμπορίου. Υπάρχουν ακόμα κάποιες λεπτομέρειες που πρέπει να οριστικοποιηθούν. Αυτό είναι υπό την ευθύνη της κυρίας Μογκερίνη, αλλά κατά κανόνα αυτό σημαίνει για την Κούβα και την εξωχώρια απόφαση των ΗΠΑ. Έχουμε εκφράσει την δυσαρέσκειά μας και είμαστε σε επαφή με τις ΗΠΑ να δούμε αν υπάρχει κάποιος τρόπος να αλλάξει η κατάσταση. Αλλά όπως ξέρετε είναι μια δύσκολη συζήτηση παρόμοια με αυτήν που γίνεται για το Ιράν. Κυρία Καβαζίνη. Ναι. Η αρχή της προφύλαξης. Είπατε ότι υπάρχουν διαφορετικές ερμηνείες. Είναι σαφές ότι υπάρχει μια σαφής αναφορά στην αρχή της προφύλαξης στην συμφωνία αυτή και ξεκάθαρη αναφορά ε, στην Συμφωνία των Παρισίων. Και ακριβώ ε, εργαστήκαμε σκληρά για να συμπεριληφθεί αυτό. Όπως ξέρετε, Υπάρχουν φήμες, υπήρχαν φήμες στην προεκλογική εκστρατεία ότι θα αποχωρούσε η Βραζιλία. Έκτοτε όμως δεν έχουν επαναληφθεί και έχουν επιβεβαιώσει ότι θα παραμείνουν στην Συμφωνία των Παρισίων και θα φροντίσουμε ε, να κάνουμε ό,τι γίνεται μέσω της συμφωνίας αυτής και άλλων επαφών για να ενθαρρύνουμε την ε, Βραζιλία να τηρήσει τις ε, δεσμεύσεις της είμαστε 100% σίγουροι ότι δεν θα μπει ε, τίποτα επικίνδυνο από τα σύνορά μας. Ποτέ δεν είμαστε 100% σίγουροι, αλλά τα κράτη-μέλη πρέπει να το ελέγχουν αυτό. Το Ρότερνταμ, παραδείγματο χάρη, είναι ένα σημαντικό σημείο εισόδου. Πολλοί κόσμοι απασχολείται εκεί σε αυτό το θέμα. Είναι ευθύνη των κρατών μελών. Προσπαθούμε να κάνουμε αξιολογήσεις κτλ κάνουν μια καλή δουλειά. Τώρα αν είμαστε 100% σίγουροι, ε, όχι. Για να είμαι ειλικρινής, όχι. Ναι, αλλά νομίζω πως κάνουν πολύ καλή δουλειά. Εάν υπάρχει κάποια ένδειξη ότι δεν δουλεύει κάτι, ε, τότε αμέσως εμείς η Γενική Διεύθυνση Ταξούντου πρέπει να αναλάβουμε δράση. Ναι, έχω Ήταν πολλές οι ερωτήσεις. Για τις είπα, κύριε Σούστερ. Όχι. Δεν υπάρχουν διαπραγματεύσεις αυτή τη στιγμή για την περιορισμένη συμφωνία για τα βιομηχανικά αγαθά. Γιατί, γιατί οι ΕΙΠΑ αναφέρονται στο κογκρέσο τους όπως έρχομαι και εγώ σε εσά και λένε δεν θα κάνουμε κάτι χωρίς τη Γεωργία και εμείς λέμε εμείς δεν έχουμε εντολή για την Γεωργία. Οπότε υπάρχει στασιμότητα. Μπορούμε να το ξεπεράσουμε, δεν ξέρω. Έχουμε δύο εντολές, όπως αντιλαμβάνεστε. Η μία ήταν για την αξιολόγηση συμμόρφωσης ε, και την εθελοντική ε, συμμόρφωση και εκεί πέρα υπάρχει κάποια πρόοδος και αυτό θα ωφελήσει εταιρείε και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού και όπως είπα ε, η έκθεση για το που βρισκόμαστε ακριβώς για τα όσα συνέβησαν από τις 25 Ιουλίου πέρσι θα δημοσιευτεί την Πέμπτη. Είναι μια μελέτη 30 σελίδων για αλουμίνιο και χάλιβα. Αυτό είναι ατυχές. Θεωρούμε λοιπόν ότι εδώ πέρα παραβιάζεται ο ΠΟΕ, η Ευρωπαϊκή Ένωση και 11 άλλε χώρες προσέφηγαν στον ΠΟΕ εναντίον των ΗΠΑ, έχουμε λάβει και αντίμετρα, έχουμε επιβάλει αντισταθμιστικά μέτρα. Αυτό είναι άτυχες, αλλά θα παραμείνουν τα μέτρα αυτά μέχρι ή, ε, όσο παραμένουν οι δασμοί γιατί θεωρούμε ότι δεν συμμορφώνονται με τον ΠΟΕ. Και επίσης πρέπει να προστατεύσουμε τη θελιβουργία μας ε, ακριβώς ε, από το dumping, ε, γιατί κλείνουν, επειδή κλείνει η αγορά των ΗΠΑ και το αξιολογούμε τώρα. Θα ληφθεί λοιπόν μια απόφαση το φθινόπωρο με πλήρη διαφάνεια πάντα. Θα σας ενημερώσουμε. Αν θα υπάρχει τώρα ομοφωνία. Ναι κύριε Κέλλη είναι μια μεικτή συμφωνία οπότε ναι θα πρέπει να υπάρξει ομοφωνία. Και να την κυρώσουν τα κοινοβούλια. Για την κατανομή των ε, ποσοστών. ναι, συνήθως είναι όποιος ε, προλάβει αυτή η αρχή ισχύει. εφαρμογή. Στην Κολομβία και στο Περού να έχουμε κάποια πρόοδο. Στην Νότια Κορέα υπάρχει κάποια διαδικασία για την κύρωση των συμβάσεων του ΑΕΛΟ. Δεν υπάρχει ακόμα πλειοψηφία στο κοινοβούλιο τους. Υπήρξε μια μεγάλη συζήτηση για το θέμα αυτό με εσά, με τα κράτη-μέλη, με τα εθνικά κοινοβούλια. Ε, και κατά βάση όλα τα μέλη ήταν κατά των κυρώσεων. Και όχι επειδή... Ε, ε, εντάξει, ακούγεται καλή ιδέα, αλλά δεν έχει βρεθεί ένα τρόπο για να λειτουργήσει. Και πρέπει άρα να είναι πολύ στοχευμένες οι κυρώσεις και χρησιμοποιείται ένα ολόκληρο φάσμα ανθρώπινων δικαιωμάτων, περιβαλλοντικών θεμάτων και εργασιακών θεμάτων. Και η συνεργασία που έχουμε με διεθνείς οργανισμούς, παραδείγματος χάνει οι ΙΠΑ προσπάθησαν να το κάνουν με τη Γουατεμάλα. Δέκα χρόνια απέτυχαν γιατί δεν μπορούσαν νομικά να αποδείξουν ότι επηρέαζε το εμπόριο, αν και υπήρχε παράβαση. Γι' αυτό επιλέξαμε αυτή τη μέθοδο. Γι' αυτό ακριβώς ε, ε, τα συζητάμε αυτά με τα μέλη εκεί να δούμε πώς ε, θα μπορέσουμε να το εφαρμόσουμε στο Μερκοσούρ θα υπάρξει μια αξιολόγηση αντικτύπου για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Θα σας την παρουσιάσουμε το συντομότερο δυνατόν, βεβαίως. Ήδη, όπως είπα, έχουμε νομοθεσία που αφορά τις υποχρέωσεις διαφάνειας για τις ευρωπαϊκές εταιρείες ε, για να αποκαλύπτουν ε, μη ε, οικονομικές προφορίες για ζητήματα εργασιακά και κλιματικά δηλαδή. Αυτό είναι ήδη η ευρωπαϊκή νομοθεσία για την αξιολόγηση. Τα μέτρα διαφύλαξη αξιολόγηση αυτών δεν ξέρω αν θα λειτουργήσει, το συζητήσαμε και προηγουμένω για τα εσπεριδοειδή. Υπόσχομαι να επανέλθω επ' αυτού μετά τις θερινές διακοπές. Μετά υπήρχε άλλη ερώτηση για το χρονοδιάγραμμα για το Βιετνάμ. Στα χέρια σας είναι αυτό. Εμείς κάναμε ό,τι μπορούσαμε. Τώρα εσείς αποφασίσετε. Νομίζω ότι αυτή η Επιτροπή με τα φιλόδοξα νέα και παλιά μέλη πρέπει να το εξετάσει χωρίς να χρονοτριβήσουμε βέβαια. Εγώ θα ήλπιζα να ψηφίσετε σχετικά σύντομα. Από σας εξαρτάται η απόφαση για την Κίνα. Πρέπει να επανέλθουμε σε μια αναλυτικότερη συζήτηση περί Κίνας στην επόμενη ε, συνεδρίασή μας. Τον Απρίλιο κουβεντιάσαμε με την Κίνα. Υπήρχε κάποια δέσμευση για τις ονομασίες προέλευσης, τις γεωγραφικές ενδείξεις. Θέλω να ολοκληρώσουμε κάτι και να συνάψουμε, ελπίζουμε, τη συμφωνία μας περί επενδύσεων του χρόνου. Σύντομα θα ξανασυντηθούμε μαζί τους και θα έρθουν σε επαφή μας για μεταρρύθμιση του ΠΟΕ για τις βιομηχανικές επιδοτήσει. τουλάχιστον είδαμε αύξηση των δεσμεύσεων και πιστεύουμε ότι η Κίνα πράγματι επιθυμεί διακαώς να διατηρήσει το πολυμερές σύστημα, διότι ωφελήθηκαν πάρα πολύ και θα χάσουν πολλά αν σταματήσει. Μπορούμε να συνεργαστούμε με τους Κινέζους εταίρους μας σε αυτό. Κύριε Ραφαέλ, δεν θα υπάρχει για τις απομακρυσμένες, τις υπερπόντιες περιοχές ε, και χτίσεις ειδική έρευνα. Θα δούμε αν κάτι έχουν κάνει υπηρεσίες μα αυτού. Δεν ξέρω. Θα επανέλθω με απάντησή μου. Δεν θα κάνουμε ειδική αξιολόγηση συνεπειών για αυτή την περιοχή. Αυτό εξαρτάται από την Ολλανδική κυβέρνηση. Μπορούμε να βοηθήσουμε βέβαια. Για τη διαφάνεια, κοιτάξτε, κάναμε πολλά. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο πλέον διαφανής διαπραγματευτεί όσον αφορά τα εμπορικά στον κόσμο. Δημοσιεύουμε αυτά που κάνουμε, συνόψει των, κάθε, των διαφόρων γύρων διαπραγματεύσεων. Έχουμε διάφορα δελτία στο διαδίκτυο, δημοσιεύουμε τι συμφωνίε από τη στιγμή που ολοκληρώνονται. Έχουμε μόνιμη συμβουλευτική ομάδα με την οποία συναντάμε τακτικά και υπηρεσίε μου ακόμη τακτικά. Και διάφοροι εμπλεκόμενοι εκφράζουν την άποψή του και δίνουν τη συμβουλή του. Ίσως μπορούμε να κάνουμε ακόμα περισσότερο, Νομίζω ότι κάναμε πολλά τα τελευταία χρόνια και ελπίζω ότι αυτό θα ακολουθηθεί από τα κράτη-μέλη να έρθουν σε επαφή με τους πολίτες τους. Και ξέρω ότι η, ΣΥΤΑ, η συμφωνία πέρασε από, τους γαλλικούς, τα γαλλικά θεσμικά όργανα και έγιναν συζητήσεις εντατικότατες όσον αφορά ε, συζήτησαν τη ΣΕΤΑ. Υπήρχαν πολλά υπέρ, πολλά κατά τα κράτη-μέλη μα δίνουν την εντολή να διαπραγματευτούμε. Εμεί δεν εμπορευόμαστε με κανένα. Το κάνουμε εκ μέρου των κρατών μελών αυτό. Τι διαπραγματεύσει. Εκπροσωπούμε τι εταιρείε οικονομία και του πολίτε των κρατών μελών. Και θέλουμε να υπάρχει και διαφανή συζήτηση με τεχνικά κοινοβούλια, περιφερειακά ε, κοινοβούλια, εμπλεκόμενου φορεί, τοπική αυτοδιοίκηση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν θα πλησιάσει του πάντε, ακόμα και αν προσπαθήσει. Αυτά. Συγγνώμη αν λησμόνησα κάτι. Α, τι είπατε. Α, κύριε Μπούτικοφερ. Η αποσύνδεση και οι γραφικές ενδείξεις Κίνα. Ναι, ελπίζω. Θα ήμασταν έτοιμοι πάνω σε αυτό με την Κίνα εδώ και καιρό. Αλλά δεν καταλήξαμε. Ο Φιλ Χόγκαν, ο φίλο και συνάδελφο, εργάζεται εντατικά πάνω σε αυτό. Ελπίζω να ολοκληρωθεί το θέμα φέτο. Αυτό αναφέρεται στα συμπεράσματα τη Συνόδου Κορυφή. Και αυτή η αποσύνδεση δεν είμαι σίγουρη ότι είναι πολύ καλή ιδέα. Ναι, μεν, συμμεριζόμαστε κάποιε επικρίσει που εκφράζουν η ΗΠΑ έναντι τη Κίνα. Δεν συμφωνούμε πάντα σε όλα. Δεν συμφωνούμε με τι μεθόδου που χρησιμοποιούνται. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να συμμορφώνεται με πολυμερεί κανόνε, να εφαρμόζει πλήρη διαφάνεια ούτω καθεξή. Δεν είμαι απόλυτα σίγουρη τι μα ζήτησαν να κάνουμε. Αλλά έτσι εκ του προχείρου θα πω ότι διστάζω. Με τα χαράς να επανέλθω όποτε θέλετε και νομίζω ότι η Σαμπίνε, η κυρία Βέιλαντ, θα είναι εδώ στην πρώτη συνεδρίασή σας μετά τις ε, θερινές διακοπές. Ευχαριστώ κυρία Πίτροπε. Με τα χαράς να σας ξαναδούμε. Θα χαρούμε να σας ξαναδούμε πριν το τέλος της ηττίας σας. Εν τω μεταξύ, ό,τι καλύτερο σε ευχόμεθα. Ευχαριστούμε πολύ. Δύσκολη αυτή η συνεδρίαση. Απαιτητική. Ελπίζω όλοι εν μέρη να έχουν ικανοποιηθεί. Σας ευχαριστώ εκ νέου. Παρακαλώ μην αποχωρήσετε. Έχω μάλλον ένα σημείο στην ημερήσια διάταξη, αρκετά γρήγορα πρέπει να είμαστε, διότι σε ένα δεκάλεπτο, 7 λεπτά θα σταματήσει η διερμηνία, οπότε θα συνεχίσουμε ανευδιερμηνία. Σα Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό καλοκαίρι. Great. So, if I may... Τέλεια. Να συνεχίσουμε λοιπόν. Έχουμε το σημείο 5 της ημερησίας διατάξεως Γενικός Προπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2020, όλα τα τμήματα. Γνωρίζετε ότι έχουμε τι... Ε, κίνηση από την Επιτροπή μας. Πρώτα απ' όλα ε, γνωμοδότηση ε, όπου αναφέρονται οι τροπολογίες και η άποψή μας, κάποιες αλλαγές στο, στα αριθμητικά στοιχεία σύμφωνα με τις επιθυμίες μας και μάλιστα οι συντονιστές αποφάσισαν ότι αυτή η γνωμοδότηση θα έχει την μορφή της επιστολής την οποία θα συγγράψει και αποστείλει ο Πρόεδρος Λάγκε. Επίσης έχουμε και τις τροπολογίες η διαδικασία ξεκινάει λοιπόν ε, και ε, λίγη η προθεσμία την 25η Ιουλίου στις 12 το μεσημέρι. Παρακαλώ λάβετε υπόψη σας ότι, το, ότι η Γραμματεία ε, θα σας μοιράσει συγκεκριμένες, συγκεκριμένα έντυπα για την υποβολή αυτών των τροπολογιών επί του προϋπολογισμού. Έχουμε μόνο πέντε λεπτάκια με διερμηνία, γι' αυτό λοιπόν προτείνω κάποια αλλαγή στο χρονοδιάγραμμα. Ίσως ε, να ακούσουμε πρώτα την παρουσίαση από την Κομισιόν, εάν υπάρχει εκπρόσωπος της Αρμοδίας Γενικής Διευθύνσεως. Uh, we can go, ε, to Α, όχι. Ωραία. Κυρία Σοφία Μουνιός, λοιπόν. Είναι εδώ. Ναι. Και μετά να ανοίξουμε τη συζήτηση η οποία θα γίνει χωρίς διαρμηνία, ε, καθότι η διαρμηνία ε, θα σταματήσει λίγη λέει ο πρόεδρος στις 5 ε, το απόγευμα η κυρία Μουνιός από τη Γενική Διεύθυνση Εμπορίου ευχαριστώ πολύ ναι, ε, εγώ είμαι από τη Γενική Διεύθυνση Εμπορίου, καθότι ε, η υπεύθυνη ε, διεύθυνση που είναι η Διεύθυνση Προϋπολογισμού δεν έχει στείλει αντιπρόσωπο σε αυτή τη στιγμή. Εν είδη εισαγωγής να σας πω ότι η Γενική Διεύθυνση Εμπορίου που συνήθως ε, στέλνει στη θέση της η Επιτροπή Προϋπολογισμού για, στη δικιά σας Επιτροπή. Δεν έχει διαφορές λοιπόν από ε, τα, τα οποία είχαν ζητηθεί προηγούμενες ε, χρονιές όσον αφορά το μέγεθος. Είμαστε μικρή γενική διεύθυνση όσον αφορά τον προϋπολογισμό, Έχουμε λειτουργικό προπολογισμό περίπου 18 εκατομμυρίων, πολύ μικρός λοιπόν, αλλά παρόλα αυτά έχουμε τη δυνατότητα με τους πόρους αυτούς να κάνουμε πολλές δραστηριότητες ε, που παρουσιάζουν ενδιαφέρον για σας, ε, καθότι το Κοινοβούλιο γνωρίζει τις δραστηριότητες μας ε, όσον αφορά την αξιολόγηση των ε, των ε, ε, εμπορικών συμφωνιών και εκ των προτέρων και εκ των υστέρων, καθώς επίσης και δραστηριότητες οι οποίες ακολουθούν την συμφωνία αλλά και την υλοποίηση της συμφωνίας. Προετοιμάζουμε σωστά την υλοποίηση των εμπορικών μας συμφωνιών και έχουμε και άλλες δραστηριότητες οι οποίες κατά κύριο λόγο σχετίζονται με το Trade Help Desk Καθώ επίση Καθώς επίσης και με κάποια άλλα εργαλεία τα οποία χρησιμοποιούμε για τη διευκόλυνση της υλοποίησης των εμπορικών συμφωνιών όσον αφορά το συγκεκριμένο προσχέδιο επί του οποίου πρέπει να γνωμοδοτήσετε, στην ουσία ζητάμε τα ίδια Ωστόσο, θα συζητήσουμε με τη Γενική Διεύθυνση Προϋπολογισμού ενδεχόμενη αύξηση αυτού του προϋπολογισμού λόγω συγκεκριμένου, ενός συγκεκριμένου ε, κειμένου της Foreign Direct Trading Proposal και για την υλοποίηση αυτού του ε, νομοθετήματος ε, συζητούμε το ενδεχόμενο αύξηση του προϋπολογισμού, το συζητούμε με τη Γενική Διεύθυνση Προϋπολογισμού. Λοιπόν, ε, μπορεί να έχουμε μικρό λειτουργικό προϋπολογισμό, αλλά δεν βασιζόμαστε μονάχα σε αυτό. Επίσης, βασιζόμαστε και σε ένα εργαλείο εξωτερικής χρηματοδότησης, είναι το Partnership Instrument, που στόχο έχει την προώθηση των ε, ε, συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όσον αφορά την πρόσβαση στην αγορά, καθώς επίσης ε, και αναπτυξιακά κεφάλαια των εμπορικών συμφωνιών. Εκεί μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε λοιπόν το κλασικό εργαλείο ε, συνεργασίας. Δεν θα πω τίποτα παραπάνω, αλλά είμαι βεβαίως στη διάθεσή σας για να απαντήσω οποιασδήποτε ερωτήσεις. Ωραία, ανταλλαγή απόψεων τώρα. Ποιος ζητάει το λόγο, παρακαλώ. Θα είμαι σύντομος. Πρώτα απ' όλα να ευχαριστούμε τον ε, Πρόεδρο Λάγκε για την ε, επιστολή η οποία νομίζω ότι ε, γενικά μπορεί να γίνει αποδεκτή. Θα υπάρξουν κάποιες μικρές τροπολογίες, τροποποίησεις τις οποίες θα σας υποβάλουμε. Σοσιαλιστέ και Δημοκράτες. Όχι. Renew. Κανείς δεν θέλει να πάρει το λόγο. Ούτε η Πράσινη, Όχι. ID. ECR. Uh, e e ο κύριος Μπουρζουάρ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Λάγκε για την ε, επιστολή. Θα ήθελα επίσης να προσθέσω κάτι στην τρίτη παράγραφο, αν είναι δυνατόν ε, εκεί όπου υπογραμμίζουμε ότι ε, χρειάζεται ενεργή δέσμευση με την κοινωνία των πολιτών και εγώ θέλω να προσθέσουμε and the stakeholders και τους εμπλεκόμενους. Δηλαδή και την κοινωνία των πολιτών, civil society, αλλά και the stakeholders ε, και τους εμπλεκόμενους. Thank you. And Gue, Mr. Gue, κύριος Yeah, want... Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και εγώ θέλω να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο. Τρεις παρατηρήσεις. Θα έλεγα ακόμα και μετά την ανταλλαγή απόψεων με την Κομισιόν να δούμε όχι μόνο τις γρήγορες διαπραγματεύσεις αλλά και χρηματοδότηση για τον έλεγχο εφαρμογής αυτών των συμφωνιών γιατί είναι ένα σημαντικό ζήτημα. Οπότε πρέπει να υπάρχουν επαρκή κονδύλια παρά την απροθυμία κάποιων κρατών μελών για την διατύπωση που λέει να διασφαλίσουμε υποφελή οικονομική ανάπτυξη. Τι είναι οικονομική ανάπτυξη. 10 χρόνια πριν η Κομισιόν μίλησε για αποανάπτυξη. Πρέπει λοιπόν να δούμε τη σημερινή κατάσταση. Δεν πρέπει να μιλάμε μόνο για ανάπτυξη, αλλά να δούμε και ζητήματα κλιματικής αλλαγής, όλα αυτά όλες αυτές τις πτυχές ε, που συζητήθηκαν και το κοινωνικό συμφέρον και τρίτον προβλέπετε κάποια χρηματοδότηση για τις ε, συμβουλευτικές αυτές ομάδες ήταν μια ερώτηση η οποία δεν έχει απαντηθεί εγώ θα επιμείνω λοιπόν ότι πρέπει να διασφαλιστεί η χρηματοδότηση γιατί η πραγματικότητα στις χώρες αυτές διαφέρει από αυτή των κρατών μελών. Σας ευχαριστώ κάποιος άλλος. Όχι. Αντίδραση από την Κομισιόν. Ναι. Να επιβεβαιώσω ότι πράγματι χρειάζεται χρηματοδότηση για την εφαρμογή των συμφωνιών αυτών και αυτό είναι κάτι βεβαίω το οποίο παρακολουθούμε με βάση τη συμφωνία. Θα φροντίσουμε να υπάρχει η χρηματοδότηση και στο μελλοντικό ενιαίο σχέσιο εξωτερικών σχέσεων οπότε βασιζόμαστε στην στήριξή σας στο μέλλον όταν θα συζητηθεί ο κανονισμός αυτός έτσι ώστε να γίνει αυτό και για τις χώριες συμβουλευτικές ομάδες όπως ξέρετε υπάρχει ένα έργο που μας επιτρέπει αυτή τη στιγμή να χρηματοδοτήσουμε τη λειτουργία αυτών των ομάδων με συμμετοχή των ειδικών και σκοπεύουμε να υπάρξει ένα ανάλογο έργο στο μέλλον, αλλά όπως είπα πρέπει να συνεχίσουμε να πιέζουμε προς το μέσο αυτό έτσι ώστε τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να συνεχίσουν να χρηματοδοτούνται. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ τελευταία παρατήρηση από τον κύριο Χάνσεν. Ήθελα να αντιδράσω σε αυτό το οποίο είπε ο κύριο Σόλτς ε, στο δεύτερο σημείο. Έχουμε βεβαίως ε, τις ε, αρχές, τις τελωνιακές. Δεν είναι αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης λοιπόν να τα κάνει αυτά. Αν δεν λειτουργεί κάτι, τα κράτη-μέλη δεν κάνουν τη δουλειά του σωστά. Εκεί κάτι πρέπει να κάνουμε σε όλα τα κράτη-μέλη για να γίνονται σωστά οι έλεγχοι. Ωραία, ευχαριστώ. Αυτά με το σημείο 5. Να σας υπενθυμίσω πως η προθεσμία τροπολογιών είναι 25η Ιουλίου το μεσημέρι. Μεθαύριο, δηλαδή. Σημείο 6. Διάφορα. Διάφορα. Όχι. 7. Επόμενη συνεδρίαση. Έχετε το χρονοδιάγραμμα μέχρι το τέλος του έτους. Οπότε η επόμενη συνεδρίασή μας είναι την Δευτέρα 2 Σεπτεμβρίου 3 η ώρα και θα συνεχιστεί και την 3η ε, Σεπτεμβρίου. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνεδρίαση.